και της Επιτροπής για το πολιετές πρόγραμμα 2010-2014 σε σχέση με το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Έχει τον λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου η κυρία Άσκ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κύριε Πρόεδρε των Επιτροπών, αγαπητοί βουλευτέ, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 και 11 Δεκεμβρίου θα εγκριθεί ένα νέο πρόγραμμα, πολιετές πρόγραμμα, για το χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας που θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα της Χάγης του 2004. Αυτό το νέο πρόγραμμα ε, ακολουθεί μια πολύ μακρά προπαρασκευαστική διαδικασία που ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια όσον αφορά μέσα στις ομάδες του μέλλοντος όπως αποκαλούνται. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και σε πολλές τοποθετήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων θέσεις της κοινωνίας των πολιτών διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία. Το πρόγραμμα είναι και αποτέλεσμα πολλών επαφών και διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βάσει της θέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικό ρόλο δημιουργώντας αυτή τη θέση και ε, έχει και νέο ρόλο το να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας. Το προγράμματα του Τάμπερε και της Χάγης αντιπροσώπευαν πάντα βήματα προόδου για την ασφάλεια, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Αλλά η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακόμα πολλές προκλήσεις που χρειάζονται λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας παρέχει νέες δυνατότητες παρέμβασης προ αυτή την κατεύθυνση. Το νέο πολιετέ πρόγραμμα, το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη, θα βασιστεί στι νέε δυνατότητε που προσφέρονται από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Το όραμα λοιπόν για το πρόγραμμα της Στοχόλμης είναι η Ευρώπη να γίνει πιο ασφαλής και να είναι και πιο ανοιχτή. Εκεί θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών. Τα δικαιώματα των πολιτών θα πρέπει να είναι η αφετηρία περισσότερο από το παρελθόν για την ε, μελλοντική συνεργασία. Εμείς θα εργαστούμε υπέρ των πολιτών και η συνεργασία στο μέλλον στην Ευρώπη πρέπει να δίνει βεβαιότητα και ασφάλεια στους πολίτες μας. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πραγματικά προβλήματα, να θέσουμε τα συγκεκριμένα ερωτήματα και να προσανατολιστούμε επί συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία μέτρα θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η συνεργασία λοιπόν σε αυτό το τομέα θα πρέπει να βασίζεται σε μια καλύτερη ισορροπία, σε μέτρα τα οποία θα πρέπει να δημιουργούν μια Ευρώπη ασφαλή και που, η οποία θα βασίζεται θα θα προχωρήσουμε βασιζόμενοι στην ασφάλεια και θα πρέπει βέβαια να προστατεύονται τα δικαιώματα του ατόμου. Η καταπολέμηση τη εγκληματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κάτι που περιμένουν οι πολίτε από την συνεργασία στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η καταπολέμηση τη διεθνού εγκληματικότητα, αλλά θα πρέπει να προστατεύονται η ελευθερία και η δικαιοσύνη. Όπω υπόθηκε και άλλη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέτρα που έχουν σαν στόχο ε, μεγαλύτερη ασφάλεια, τα μέτρα που δίνουν ε, παρέχουν δικαιοσύνη και εγγυώνται την επικράτηση του κράτους δικαίου θα πρέπει να προχωρούν όλα μαζί ταυτόχρονα ισότιμα. Θα πρέπει να είναι πραγματική δυνατότητα. Όσον αφορά την καταπολέμηση διεθνού εγκληματικότητα, έχουμε τεράστιε προκλήσει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε το εμπόριο ναρκωτικών, το εμπόριο των ανθρώπων, τρομοκρατία. Είναι μια πραγματικότητα στην Ήπειρό μα. Έχουμε νέε μορφέ εγκληματικότητα, παραδείγματο χάρη αυτή που βλέπουμε και στο διαδίκτυο δεν ε, μπορούμε ε, να τα αφήσουμε έτσι τα πράγματα. Τα σύνορα ε, να εμποδίζουν τις αρχές που καταπολεμούν την εγκληματικότητα και να εμποδίζονται από τα σύνορα. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί αυτή. Αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε για να έχουμε συνεργασία αστυνομική και σε θέματα ποινική δίωξη στην Ευρώπη. Πρέπει να βρούμε κοινέ λύσει στα κοινά προβλήματα. Μία συνεργασία σε αστυνομικό επίπεδο, μία καλή ανταλλαγή πληροφοριών και μέθοδοι εργασία ανεπτυγμένε αντιπροσωπεύουν τη βάση για να χειριστούμε αυτά τα προβλήματα. Ένα σημαντικό τμήμα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος από πλευράς της ένομης τάξης είναι και η αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχουν τυποποιημένες τέτοιες διαδικασίες που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες για την ανταλλαγή πληροφοριών. Έχει τεράστια σημασία επίσης να διασφαλίζουμε ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών, αυτή η ροή πληροφοριών θα υλοποιεί όλους τους αναγκαίους στόχους, όπως για παράδειγμα την, τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και των στοιχείων αυτής της ιδιωτικής ζωής, προσωπικών δεδομένων και όσον αφορά τράπεζες δεδομένων ε, δεν θα παραβιάζουν αυτές τις αρχές. Πρέπει να δημιουργηθεί η Ευρώπη της ασφάλειας με αυτή τη βάση, όπου το έγκλημα θα καταπολεμάται αποτελεσματικά, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών θα προστατεύονται και θα διασφαλίζονται. Είναι αναγκαίο και τα δύο διτά να γίνουν. Πρέπει να υπάρχει η σωστή ισορροπία ισορροπία στις δράσεις που θα επιλέγονται πάντα. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ένα ουσιαστικό συστατικό στοιχείο για αυτού του είδους τη συνεργασία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να, κατα... να επιτυγχάνουν τις αποφάσεις και την ομολογία άλλων κρατών μελών να τις αναγνωρίζουν και να τις εκτελούν. Αυτό προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Πρόκειται για την ίδια την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατικών αρχών των χωρών μελών μας, αλλά και οι ίδιοι οι να μπορούν να αισθάνονται εμπιστοσύνη όταν τέτοια σημαντικά μέτρα αποφασίζονται από εμά. Μία οδό, ένα τρόπο για να αυξηθεί αυτή η εμπιστοσύνη είναι η αύξηση, η αναβάθμιση του επίπεδου ε, στοιχείων και γνώσεων και αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύωση, μέσω δικτύων, μέσω ε, μηχανισμών ε, σωστή αξιολόγηση σε διαδικτύωση. Όταν πρόκειται για την προαγωγή τη εμπιστοσύνη πρέπει να διασφαλίζουμε ότι οπουδήποτε χρειάζονται αυτέ οι δράσει. θα διασφαλίσουν τους πολίτες παντού. Πρόκειται για απλά πράγματα, απλές, απλές διαδικασίες, χρήση μιας γλώσσας που θα είναι εύληπτη και κατανοητή για τους κατηγορούμενους, τους εναγόμενους για παράδειγμα, ή ποια είναι τα δικαιώματα κάποιου που θεωρείται ύποπτος ή είναι θύμα μιας διαδικασίας. Είναι είναι το ότι υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας για ένα τέτοιο δρομολόγιο, για ένα τέτοιο πρόγραμμα από πλευρά του Συμβουλίου όταν υπάρχουν υποψίες ή πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι ένα και στις διαδικασίες αυτών να αποτελέσει και ένα τμήμα του προγράμματος της Στοχόλμης. Ελπίζω ότι θα επιτευχθεί αυτό. Το πρόγραμμα της Στοχόλμης επίσης θα δίνει μια ε, σαφή προοπτική υπέρ των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Θα πρέπει από πλευρά των άλλων κρατών μελών να συντάσσονται οι πληροφορίες και τα στοιχεία σε μια εύληπτη γλώσσα, να υπάρχει υποστήριξη ώστε να υπάρχει πληροφόρηση και ενημέρωση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια δίκη, ώστε τα θύματα να μπορούν να την χάνουν και αποζημίωση ε, για την ε, απώλεια δικαιωμάτων τους. Ε, επίσης κάποια θέματα όσον αφορά νομικά ζητήματα που σε πολύ μεγάλο βαθμό φυσικά αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών άμεσα. Ένα συγκεκριμένο τέτοιο ζήτημα είναι η επεξεργασία του κανονισμού Βρυξελών ε, υπαριθμών 1 για το τι θα γίνεται από τα κράτη-μέλη. Ίσως ακούγεται πολύ τεχνικής φύσεως αυτό το θέμα, όμως αφορά τους πολίτες της Ένωσης ε, με ιδιαίτερο τρόπο. Ένα άλλο θέμα είναι η κατάργηση της, ε, της διαδικασίας εξεκβάτων. Πρέπει δηλαδή η διαδικασία αυτή, όπως προέβλεπε, να υποβάλει αίτηση σε ένα κράτος μέλος ε, και μετά από έγκριση αυτού του κράτους μέλους να εξετάζεται η δυνατότητα δίκης και η δυνατότητα κατάργησης αυτής της διαδικασίας πρέπει να βαίνει παραλλήλου με την η διασφάλιση ε, ε, δικαστικών εχεγγύων και ρητρών ασφαλείας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το ότι μπόρεσε να γίνει λόγος για αυτό το θέμα ε, σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στο να ακούσω τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Είμαι στη διάθεσή σας για την απάντηση ενδεχομένως ερωτήσεων. θα ήθελα να δώσω τον λόγο και στη συνέχεια για αυτά τα θέματα στον συνάδελφο που είναι αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Σημαντικά ζητήματα και για την ε, μελλοντική αυτή συμφωνία της Στοκχόλμης. Παρακαλώ. Äh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια πολύ καλή θετική συνεργασία όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γραφείο υποστήριξη για θέματα ασύλου. Υπάρχουν κάποια τυπικά θέματα που εκκρεμούν ακόμα και πρέπει να επιληθούν, όμω δημιουργήθηκαν οι προποθέσει ω βάθρα για τη λειτουργία αυτού του γραφείου. Με πολύ θετικό πνεύμα αντιμετωπίζει αυτό το θέμα συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο, διότι ότι καταφέραμε να πετύχουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα και είναι ένα καλό μήνυμα για την περαιτέρω συνεργασία που υπό το φως της έναρξης ε, της λειτουργίας της συνθήκης Λισαβόνας θα πρέπει να λειτουργεί. Ταχεία λήψη αποφάσεων ε, σε σχέση με αυτό το γραφείο είναι ένα καλό παράδειγμα, μια καλή συνεισφορά για αποτελεσματική διαμόρφωση των δικαιωμάτων συναπόφασης. Αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα είναι το επόμενο πενταετές πρόγραμμα για τον τομέα δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων. Θέλω καταρχήν να πω ότι πολλά έχουν γίνει Πολλά έχουν γίνει ήδη κατά το παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το άσυλο και τη μετανάστευση. Λάβαμε αποφάσεις για παράδειγμα, για μια κοινή νομοθετική προσπάθεια και κοινό νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να έχουμε μια κοινή μεταναστευτική πολιτική ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα κοινό σύστημα για τη χορήγηση ασύλου. Και αντιμετώπιση παρόμοιων θεμάτων. Είχαμε και το πρόγραμμα του Τάμπα και το πρόγραμμα της Χάγης στο παρελθόν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά το παρελθόν έτο, συνήψε το σύμφωνο για το, τη μετανάστευση και το άσυλο. Και πολλές προσπάθειες έγιναν και μεγάλο έργο ε, επετελέστη. Τώρα είναι η χρονική στιγμή για τη συνέχιση αυτών των πολιτικών με ένα, σε ένα νέο πλαίσιο. Το σημείο φετηρίας πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια χρηστή διαχείριση ω ως ε, ε, πολιτική από πλευρά μας για τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης, για τα κράτη-μέλη αλλά και για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, για τις χώρες προέλευσης των μεταναστών και τους επιμέρους ετούντες άσυλο ή και μετανάστες. Αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο, η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια δυναμική ανταγωνιστική περιοχή του κόσμου, τότε θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα πράγματα, να ρυθμίσουμε τη μετανάστευση περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, να ρυθμίσουμε αυτά τα πράγματα υπό το φως κιόλα και των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για να τονίσουμε τη διεθνή αυτή διάσταση, το θέμα τη συνεργασία με τι χώρε προέλευση και διαμετακόμιση και χώρε διέλευση δηλαδή, η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ε, διαμόρφωση του προγράμματο τη Στοχόλμη. Θα πρέπει εδώ να παγιωθούν ε, τα πρώτα βήματα που έγιναν και η συνεργασία, ε, η συνάρτηση μεταξύ και μετανάστευση, αυτή η συνάφεια και συνάρτηση πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από πλευράς μας μοχλό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Διαπιστώθηκε κατά το παρελθόν ότι τα κράτη-μέλη εδώ από κοινού προτίθενται να καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαμορφώσουν μια σωστή πολιτική παλινόστηση ή επιστροφής των ατόμων αυτών στις χώρες τους. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Frontex ως υπηρεσία έχει ε, σημαντικό ρόλο να επιτελέσει και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβούν σε μια ενδυνάμωση, τόνωση των δραστηριοτήτων της Frontex ε, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Εδώ η συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και τις χώρες προέλευσης αυτών των μεταναστών, αυτών των ατόμων είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Είναι σημαντικό το θέμα στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Πρέπει να αναζητήσουμε τη σωστή ισορροπία ώστε τα μέτρα τα οποία θα υιοθετηθούν να μην αποβούν εις ε, μιας και να μην δημιουργούν προσκόμματα και επιβάρυνση στην ε, μεταναστευτική μας πολιτική ή στους ε, άσυλο που μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται θέτουν έτοιμα χωρίσεις ασύλου. Θα πρέπει να προστατευτούν ε, οι, ομάδες, οι ευάλωτες ομάδες και τα ασυνόδευτα παιδιά ή τα ανήλικα παιδιά και το θέμα της αλληλεγγύης και της επιμεριζόμενης ευθύνη είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρουμε στο πρόγραμμα στο Στοχόλμης. Δεν υπάρχουν απλές λύσεις. δράση μας πρέπει να, να είναι στις δράσει μας να μπορέσουμε να βασιζόμαστε σε ευρύτερη βάση για να ρυθμίζονται αυτά τα θέματα. Μία συνεργασία με τρίτες χώρες διαδραματίζει σημαντικό παράγοντα εδώ. Ένα είδος μηχανισμού αλληλεγγύης με άλλα λόγια για την υποστήριξη εκείνων των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη επιβάρυνση και που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό τέτοιων μεταναστών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να τύχουν ακριβώς την υποστήριξη των υπόλοιπων και την, αλληλεγγύη των υπόλοιπων κρατών μελών. Η Frontex πρέπει να έχει σημαντικότερο ρόλο στην στην επιστροφή, επανεισδοχή τέτοιων ε, μεταναστών. Στόχο πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενό μηχανισμού συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών αλλά και, μεταξύ, και με τρίτες χώρε Πρέπει να είναι σαφέ ότι εδώ συνολικές δράσεις ε, που θα καλύπτουν το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούνται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Σημαντικό είναι το πρόγραμμα τη Στοκχόλμης να υλοποιεί αυτού του στόχου. Ένα κοινό δηλαδή μεταναστευτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα για τη μετανάστευση μέχρι το 2012. Θα, μέχρι το 2010, με συγχωρείτε. Πρέπει να είναι σαφές ότι θα έχουμε μια αποδοχή αυτού του προγράμματος και οι όσοι θα ε, εμπλέκονται να εντάσσονται στα κριτήρια αυτά ανακράτος μέλος στα οποία θα εφαρμόζονται οι αρχές αυτές φυσικά χρειαζόμαστε μια πολύ καλή συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο. Εδώ τα θέματα χωρίσης ασύλου αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τμήμα. Ένας άλλος σημαντικός πυλώνας αυτού του, αυτής της προσέγγισης είναι η εξωτερική διάσταση κυρίως με την εγκατάσταση ε, προσφύγων από τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα υπέβαλε μια πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή νέα πολιτική μετεγκατάστασης ή εγκατάστασης ε, προσφύγων προσφύγων. Υπό αυτό το πρίσμα ε, κάποια κράτη-μέλη που θέλουν να αντανακλώνται αυτές οι αρχές στο πρόγραμμα της ε, Στοχόλμη για να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα χωρίς ασύλου μέχρι το 2012, όμως για να γίνει αυτό το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεργάζονται πολύ στενά. Λοιπόν, θα πρέπει ε, να θεθούν προτάσει νομικέ επιτάπητο και θα πρέπει τελικά αυτέ να εφαρμοστούν οι σωστέ προτάσει. Μετά, έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνδέεται με το εσωτερικό έργο των κρατών μελών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα πρόοδο, όχι μόνο στα πλαίσια τη ε, πολιτική ασύλου και μεταναστευσεω, διότι είμαστε ένα φορέα ε, παγκόσμια εμβέλεια. Δεν θα πρέπει ποτέ να αποκρύπτουμε τη συνεργασία που πρέπει να έχουμε με τις τρίτες χώρες. Διότι ε, γνωρίζουμε ότι και εξωτερικές σχέσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο. Λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές γραμμές της προτάσεως του Συμβουλίου όσον αφορά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Είμαστε στο τέλος μιας μακράς περίοδου διαπραγματεύσεων και ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα θα μπορέσει να υιοθετηθεί ε, μέσα σε λίγες εβδομάδες. Τώρα, εν συντομία, να δούμε κάποιες πτυχές που αφορούν τη συνθήκη της Αβώνας. Η νέα συνθήκη της Αβώνας επιφέρει πολλές καινοτομίες στον τομέα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θα έχουμε λοιπόν την διαδικασία, την νομοθετική, την κανονική νομοθετική διαδικασία, συνηθισμένη νομοθετική διαδικασία που εισάγεται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή θα έχει ενισχυμένο ρόλο να διαδραματίσει στην νομοθετική αυτή διαδικασία. Μαζί με την ε, Υπουργό ΑΣΚ θέλουμε να έχουμε πιο ενισχυμένη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν νέα καθήκοντα και αυτό θα μπορέσει να ενισχύσει το δημοκρατικό έλεγχο όσον αφορά αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ όπως και η συνάδελφός μου η Μπέτε Σάσκ ε, διότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη συζήτηση και να δώσουμε απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπίλστρο. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λάβει τον λόγο ο Επίτροπος Μπαρό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε μετά από τις έξοχες παρουσιάσεις της Μπεατρίς Άσκ και του Τομπίας Ρίλστρομ θα ήθελα, για να παραμείνω στα ουσιώδη, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία η οποία στην ανακοίνωσή της διαφύλαξε το πνεύμα του προγράμματος της Στοκχόλμης και έθεσε τον πολίτη στο επίκεντρο της δράσεως. Ελπίζουμε αυτό το κείμενο που θα πρέπει να εθετηθεί στο επόμενο Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνη και μετά θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου αυτό το κείμενο να είναι φιλόδοξο, ισορροπημένο και προφανώς να αντικατοπτρίζει τις νέες θεσμικές ισορροπίες. Τώρα θα είσαστε συνομοθέτες σχεδόν σε όλους ε, τους τομείς του θεμάτων εσωτερικών και ασφαλείας και δικαιοσύνης και αυτή η κοινοβουλευτική χρειά που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψους αποφάσεων, επίσης μεγαλύτερο έλεγχο από τα εθνικά κοινοβούλια και τις διάφορες εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό για τον μεγάλο αυτό χώρο της ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας είναι μια ευκαιρία. Είναι πολύ καλό που συμμετέχουν τα κοινοβούλια σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα έρχομαι στις προτεραιότητες που υπογραμμίσατε στο σχέδιο ψηφίσματός σας. Τονίζετε το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σωστά επιμένετε επί της ελεύθερης διακίνησης ε, που είναι μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο προφανώς δεν πρέπει να υπονομεύεται και να αμφισβητείται. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε δύο τομείς προόδου σημαντικές. Η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων γίνεται δεσμευτική και άνοιξε ο δρόμος για την προσχώρηση της ενώσεως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως υπογραμμίζεται στο ψήφισμά σας, πρέπει να έχουμε ένα πλήρες καθεστώς προστασίας δεδομένων, να καταλήξουμε εκεί, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές ε, εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μία ανακοίνωση το 2010 πάνω σε αυτό το θέμα. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να καλύψουμε όλες τις πολιτικές της ενώσεως με αυτό το πλήρες καθεστώς της προστασίας των δεδομένων. Επιμένετε επί της προστασίας των παιδιών και με τη Σουηδική Προεδρία ε, ε, ε την Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού διότι ήταν η 20η επέτειος αυτής. Θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή οσον αφορα αυτα τα θεματα ευρωπαικη ενωση και γι' αυτό θα υποβάλουμε ένα σχέδιο δράσος όσον αφορά τους, τα μη συνοδευμένα ανήλικα παιδιά αρχές του 2010. Εν γέννη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θέλουν τα ίδια όσον αφορά την καταπολέμηση κάθε διάκρισης και όσον αφορά την προώθηση ισότητας ανδρών και γυναικών και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούν στην προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο των δράσεων τον πολίτη. Ελεύθερη διακίνηση, εκλογικά δικαιώματα, ε, προξενική προστασία. Θα μπορέσουμε τώρα όλα αυτά ε, να τα εφαρμόσουμε. Η συνθήκη της ε, Λισαβόνας δικαιώνει, δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να κινούνται και ε, θα εκδώσουμε πράσινη βίβλο πάνω σε αυτό το θέμα και θα υποβάλουμε πρόταση το 2010 βάσει των διαβουλεύσεων που θα λάβουν χώρα. Όπως είπε πάρα πολύ καλά η κυρία Υπουργός, η Μπεατρίς Άσκ, χρειαζόμαστε οι δικαστές των κρατών μελών να έχουμε μια ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα κοινή. Πώς, μέσω της κατάρτισης μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης αναλάβαμε μια δέσμευση. Τουλάχιστον οι μισοί δικαστές και οι εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει μια ευρωπαϊκή κατάρτιση ή να έχουν συμμετάσχει σε μια ανταλλαγή συναδέλφους τους από άλλο κράτος. Υπογραμμίζεται επίσης την ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και υποστήριξη της εύρυθμης ε, λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τονίζεται την προστασία των θυμάτων. Θυμάτων οικογενειακής βίας, ε, θυμάτων τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επ' αυτών των θεμάτων θα υποβάλει πρόταση δρατώμενοι των ευκαιριών που παρέχει ε, η συνθήκη της Αβώνας. Όσον αφορά την πτυχή ε, προστασία και ασφάλεια υπογραμμίζεται την έλλειψη γενικής στρατηγικής όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων και την ε, δομή της ασφαλείας. Όπως είπε πολύ καλά και η κυρία Μπεατρίς Άσκ, γι' αυτό το πρόγραμμα της Στοχόλμης εμπεριέχει πραγματική στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας στρατηγική που ε, συμμορφώνεται με τις επιταγές των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμπληρώνει την στρατηγική για την εξωτερική ασφάλεια. Αυτή η γενική στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας εδράζεται επί συνεργασίας όσον αφορά αστυνομικά θέματα και θέματα ποινική δικαιοσύνης και όσον αφορά τη διαχείριση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Όπως εξηγήθηκε πάρα πολύ καλά από τον κ. Τομπίας Μπίλστρομ, η πολιτική μετανάστευση θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο και όραμα για βελτιστοποίηση της συνεισφοράς της μετανάστευσης στο κοινωνικό, ε, στο κοινωνικό και οικονομικό τομέα και τις εξελίξεις. Θα πρέπει να είναι σαφές το πλαίσιο για τους νόμιμους μετανάστες και να τους δοθεί το σωστό καθεστώς θα πρέπει να μειωθεί και να προλαμβάνεται η παράνομη μετανάστευση με σεβασμό στα ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα τα ανθρώπινα. Περιγράφουμε σε αυτό το τμήμα ποια είναι η γενική προσέγγιση που επιτρέπει να συνδέουμε ανάπτυξη και μετανάστευση. Όσον αφορά άσυλο. Όσον αφορά το άσυλο λοιπόν, συνυπογράφω την έκκλησή σας για μια ειλικρινή αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών. Η Ένωση θα πρέπει να καταστεί ένας πραγματικός χώρος, αλληλέγγυος χώρος προστασίας επί τη βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τα πρότυπα προστασίας και όπως λέει ο κύριος Μπίρστομ, το άσυλο θα πρέπει να δίδεται επί τη βάση ιδίων κριτηρίων απαιτείται αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών και ιδιαίτερως ε, οι χώρες εκείνες οι οποίες δέχονται ε, ροή ε, μεταναστών ή προσφύγων. Τώρα, ως προς τον χώρο ασφάλειας και δικαιοσύνης. Υπάρχει μια εξωτερική διάσταση ισχυρή και απόλυτα συνεπής με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται στο ψήφισμά σας επανειλημμένως τη σημασία του, της επιτήρησης, της εποπτείας και της αξιολόγησης. Στο σημείο αυτό συμμεριζόμαστε και εμείς την άποψή σας. Θα πρέπει να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των πολιτικών και των προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ε, τεθούν σε εφαρμογή και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε τις πιθανές επιπτώσεις ε, επί των ε, πολιτών και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν τα απαραίτητα μέσα. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για την υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης. Τονίζω την ικανοποίησή μας για την ε, καλή συνεργασία με τη Σουηδική Προεδρία με την οποία κάναμε μια, ένα πολύ σοβαρό έργο και η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική για μας αυτές τις τελευταίες στιγμές που μας χωρίζουν από την υιοθέτηση του προγράμματος της Στοκχόλμης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γι' αυτό ακριβώς σας ευχαριστώ θερμά και με τη σειρά μου θα σας ακούσω με μεγάλη προσοχή. Σας ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Περνάμε στην ομάδα παρεμβάσεων των κοινοβουλευτικών ομάδων για το ΕΛΚ. Θα λάβει τον λόγο για δύο λεπτά ο παρακαλώ. Κύριος Βέμπερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι εδώ και πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζομαι στον τομέα εσωτερικών υποθέσεων και των νομικών θεμάτων. Είναι χαρά για μένα όταν για τα επόμενα χρόνια μπορούμε να έχουμε συνομοθετική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Χρειαζόμαστε αυτό το χαρτοφυλάκιο που να κινεί και να συγκινεί τους πολίτες. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και ζητούν οι πολίτες, προκαλούν και ζητούν απαντήσεις από εμάς. Γι' αυτό θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ στις αλλαγές που απορρέουν από τα νέα νέα βάθρα, νέε βάσει εργασία που θα έχουμε και τα θέματα, θεματολογικά. Συνεργασία με το Συμβούλιο. Έχουμε εκπροσώπους του Συμβουλίου που λένε εδώ πολλέ φορέ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ότι είναι σημαντικό το θέμα συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ πολλέ φορέ ε, δεν ανταποκρίνονται απόλυτα. Είναι δική μα δουλειά ω ε, ε, ευρωβουλευτέ να ζητούμε από το Κοινοβούλιο να λαμβάνονται υπόψη αυτέ οι αρμοδιότητε μα. Μελλοντικά δεν θα είναι πλέον, δεν θα απουσιάζει το θέμα της συναρμοδιότητας και συνομοθεσίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι δεν θα μπορούν πλέον να μας αγνοούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να δίνουμε ιδέες εμείς ως Ευρωβουλή. Έχουμε την ευκαιρία με τη νέα συνθήκη να υποβάλουμε πρωτοβουλίες. Ιδέες για πρωτοβουλία και ανάληψη πρωτοβουλειών. Πρέπει να έχουμε, θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα μελλοντικά να δρούμε ως συνομοθέτης και προ, υποβάλλοντας προτάσεις και πρωτοβουλίε. Πρέπει να είμαστε και εταίροι όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, ε, Παράνομη μετανάστευση. Όχι μόνο να έχουμε τι θέσει των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά να είμαστε σοβαρό εταίρο. Και το θέμα τη επικουρικότητας πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από την Ευρωβουλή. Όταν θα είμαστε υπεύθυνοι πρέπει να αντανακλώνται με τον καλύτερο τρόπο σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσει, περιφερειακά, ευρωπαϊκά ή ε, αναχώρα. Έχω τους, αυτές, αυτούς τους άξονες που θα ήθελα να ληφθούν υπόψη με το πρόγραμμα τη Στοχόλμης ε, ενισχυμένα. Αυτή η φάση όμως είναι φάση ικανοποίηση που πρέπει να εκφράσουμε και θα στραφούμε στην εργασία, στη δουλειά μα, ανασκουμποθούμε και θα δουλέψουμε καλά. Σα ευχαριστώ για τη σοσιαλιστική ομάδα για ένα λεπτό. Η κυρία Φλασικόβα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ένα πολύ σημαντικό βήμα γίνεται για την επιτυχία ε, αυτού του εγχειρήματο είναι η έγκριση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Η διαδικασία τη συνθήκη τη Λισαβόνα θα ενισχύσει από εκ των έσω την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα ενισχυθούν και οι σχέσει προ τα έξω και θα υπάρχει συνεργασία στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα. Θα είναι πιο ανοιχτή και πιο αποτελεσματική, πιο δημοκρατική ένωση. Βασική πρόκληση και βασική προτεραιότητα είναι να διαφυλάξουμε τα βασικά δικαιώματα και τι βασικέ ευθύνε, καθώ και την ακαιρεότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη μέσω τη υποστηρίξεω πλήρου εφαρμογή και τελείου σεβασμού και βελτιώσεω των νομικών μέσων που υφίστανται για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ε, ε, ευθυνών των πολιτών. Η διαδικασία τη Στοχόλμη υπογραμμίζει τα δικαιώματα και στον τομέα τη ασφαλεία και τη δικαιοσύνη. Θα πρέπει αυτού του μηχανισμού να εκμεταλλευτούμε για τη βελτίωση πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να βελτιώσουμε και την αποτελεσματικότητα τη απονομή τη δικαιοσύνη σε όλη την Ευρώπη και την εφαρμογή του κράτου δικαίου σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να βελτιωθεί η αστυνομική συνεργασία και να βελτιωθεί η ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη. Τι ο τρόπο θα πετύχουν του στόχου. Θα ευχαριστήσω όλου του ηγητέ και ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε, κύριε Φλασικόβα. Για του φιλελεύθερου δημοκράτε θα λάβει τον λόγο για δύο λεπτά η κυρία Χένισε Φλασάρτ, παρακαλώ. Thank you very much. Well... Ευχαριστώ. Μπορώ τώρα να συνοψίσω ε, πάρα πολύ σύντομα το ψήφισμα των 27 σελίδων, αλλά δεν θα το πράξω. Απλώς θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία. Σε μια πτήση της ε, British Airways από το Johannesburg, μια γυραιά κυρία κάθεται ε, δίπλα σε έναν ε, μαύρο. Λέει, ζητάει λοιπόν να της αλλάξουν τη θέση. Λίγα λεπτά αργότερα έρχεται η αεροσυνοδός και της λέει «Κυρία μου, δυστυχώς η, η οικόνομη είναι πλήρης». Μίλησα με την υπεύθυνη και η διακεκριμένη θέση είναι και αυτή πλήρης. Έχουμε όμως μία θέση στην ε, πρώτη θέση, στην και είναι πάρα πολύ σπάνιο να κάνουμε τέτοια αναβάθμιση. Το Γεγονός όμως ότι έπρεπε η κυρία οπωσδήποτε να αλλάξει θέση έρχεται και λέει στον κύριο Κύριε, μπορείτε να πάρετε τα πράγματά σας και να περάσετε στην πρώτη θέση και να καθίσετε εκεί. Οι άνθρωποι που κάθονταν γύρω από τους επιβάτες άρχισαν να χειροκροτούν. Αυτά όλα τι σχέση έχουμε εμάς θεωρούμε τους άλλους κατώτερους από εμά. Η λευκή νοτιοαφρικανική, νοτιοαφρικανή κυρία έτσι αισθανόταν. Ωστόσο, κάποιοι συνάδελφοι από το ΕΛΚΑ αλλά και από το Συμβούλιο κατανοούν απολύτως αυτό που προσπαθώ να πω. Η δική μου ομάδα, η ΑΛΤΕ, πιστεύει ακράδαντα ότι οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν να κατανοήσουν και να εμπιστευθούν την Ευρώπη. Μια τέτοια Ευρώπη θα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι θεμελιώδει αρχέ, τη δημοκρατία, την ένωμη τάξη και βεβαίως την ισότητα για όλους. Είναι καιρό λοιπόν να εξαλείψουμε κάθε μορφή ε, διάκρισης και και τις διακρίσεις εκείνες που έχουν ε, ε, να κάνουν με τη διαφορά του φύλου. Σας ευχαριστούμε για τους πρασίνους και την Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τρία λεπτά. Ο κύριος Άλμπρεχτ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαρωτόμαστε σοβαρά πώς μπορεί να γίνεται εδώ με ένα ψήφισμα για να αποφασίζουμε για ένα παλαιότατο πρόγραμμα. Διότι εχθές μόλις η, Ευρωπαϊ... η Προεδρία του Συμβουλίου, η Σουηδική Προεδρία υπέβαλε νέο πρόγραμμα Υποθέτω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του σώματος δεν μπόρεσε αυτό το σχέδιο να το διαβάσει ακόμα. Αυτό είναι νομίζω κάτι απαράδεκτο ως κατάσταση ε, και μελλοντικά κιόλα ε, μέσα στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο η διαδικασία που οδήγησε σε αυτό το ψήφισμα είναι, ήταν ε, μη διαφανής και εν μέρη χαοτική. Οι μικρές ομάδες είχαν αποκλειστεί από τις διεργασίες και μια ολόκληρη σειρά τροπολογιών σε σχέση με την λήψη απόφασης με δημοκρατικό τρόπο την δυσχέρανε σοβαρά. Γι' αυτό δείξτε κατανόηση και συγχωρέστε μας που ζητάμε ξεχωριστή ψηφοφορία σε πολλά θέματα. Split votes. Το Κοινοβούλιο πρέπει σε βάθος να προβληματιστεί και να δει και έναντι του Συμβουλίου και μέσα στο ίδιο το Κοινοβούλιο πώς θα αντιμετωπίζει τέτοια θέματα. Για το περιεχόμενο του προγράμματος της Στοχόλμης. Αδιαμφισβήτητο είναι ότι τμήματα, μέρη αυτού του προγράμματος είναι πρόοδος, αυθεντική πρόοδος στον τομέα τη δικαιοσύνη και για την ε, κατάρτιση και επιμόρφωση βλέπουμε να υπάρχει ένα θετικό σημείο ως αφετηρία για τα επόμενα χρόνια. Όμως, σε σχέση με το συσχετισμό των πολιτών προς το κράτος, αυτό το πρόγραμμα είναι, αν θέλετε, μία ε, εκδήλωση, μία δήλωση λανθασμένων προθέσεων. Και στην πολιτική ασύλου και στην πολιτική ε, ολοκλήρωσης και στην προστασία προσωπικών δεδομένων η απέτηση για ασφάλεια στην Ευρώπη πριτανεύει και θεωρούνται επουσιοδέστερα θέματα οι ιδιωτικές ελευθερίες ε, και τα θέματα πολιτικών ελευθεριών. Διαρωτώ με, πού βρίσκεται εδώ η ιδέα, της, ε, η ιδρυτική ιδέα, ο μύθος που είχε δημιουργηθεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δημιουργούνται φοβίες ε, και αναζωπυρώνονται φόβοι και φοβίες. Και σε σχέση με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, όχι μόνο για αυτό, αλλά φοβίες στους πολίτες της Ευρώπης για εκείνους που θέλουν να έρθουν ως μετανάστες στην Ευρώπη και να μείνουν ανάμεσά μας. Και δυσχεραίνονται τα πράγματα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και δυστυχώς και με με το ε, κείμενο της πρότασης ψηφίσματος ε, υπάρχει διασύνδεση εσωτερικής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής. Εποπτεία και παρακολούθηση όλων των πολιτών στην Ευρώπη και παρακολούθηση και ενίσχυση των δράσεων της Frontex. Πρέπει η Ευρώπη να απόσχει από αυτή την τάση και να ε, θέσει τα θέματα σε, ένα μια σωστότερη βάση. τελευταία, ακροτελεύτια παρατήρηση. Και εδώ θα, ήθελα να πω ότι θα πρέπει οι πολίτες να είναι ε, υπεύθυνοι σε σχέση με τις τοποθετήσεις ε, όταν για παράδειγμα πώς θα αντιμετωπιστούν τα θέματα της συμφωνίας SWIFT. Γιατί στα θέματα της πολιτικής ασφάλειας όπως η συμφωνία SWIFT πάλι εκ νέου υπαναχωρούμε εναντί των ΗΠΑ και των απαιτήσεών τους χωρίς να υπάρχει σε βάθος συζήτηση. Και γιατί από το Συμβούλιο διαρκώς και διαρκώς ως Κοινοβούλιο ε, αφήνουμε να χειραγωγούμεθα και να αποκλίνουμε από τις προθέσεις μας. Εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες εδώ και τώρα για τις πολιτικές ελευθερίες και θα πρέπει εδώ να υπερψηφίσετε τις τροπολογίες μας. Έτσι εμείς ε, ως πράσινοι αν δεν γίνει αυτό δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την πρόταση ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Άλμπρεχτ. Στη συνέχεια για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές για δύο λεπτά θα λάβει τον λόγο ο κύριος Κέρκχοπ. Προεδρέ, Επίτροπε, η πρόταση ψηφίσματος που συζητούμε είναι τέλειο παράδειγμα πρέπει να πω τη χειρότερη εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παραδέχομαι ότι οι συγγητέ εργάστηκαν σκληρά, είχαν πολύ αξιέπαινε προθέσει, προσπάθησαν να συμπεριλάβουν τα πάντα σε ένα κείμενο 27 σελίδων. Είναι συγκεχημένο το κείμενο, κατά απόψη μου, και πολύ λιγότερο. Δεν έχει την αξία που δεν είναι αυτό που θα άξιζε η Σουηδική Προεδρία και το πρόγραμμα τη Στοχόλμη. Θέλουμε να συμβάλλουμε στο να βρούμε λύσει και να υπάρχει αλληλεγγύη όσον αφορά την καταπολίτευση διαφορά και αντιμετώπιση τη μετανάστευση και ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά όμω δεν θα πρέπει να γίνουν ει βάρο εθνική κυριαρχία, ούτε θα πρέπει να είναι πολύ περιοριστική όρη που θέτουμε. Εάν εφαρμόσουμε τη Σύμβαση 1959 του ΟΗΕ, τη Σύμβαση για του Πρόσφυγε, σωστά, ε, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα σύλλου. Και υποστηρίζουμε ανταλλαγή πληροφοριών, να εξασφαλίσουμε το ότι έχουμε πραγματική προσέγγιση για ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια χώρου δικαιοσύνη και να υπάρχει ισχυρή προστασία των δεδομένων, αλλά καταναλογικότητα, αναγκαιότητα και διαφάνεια. Βάσει αυτών των αρχών υποστηρίζουμε επίση την αρχή τη αμοιβέ αναγνωρίσεω και ελεύθερη διακίνηση. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να κινούνται ελεύθερα. Η κατάχρηση των δικαιωμάτων όμω πρέπει να περιορίζεται μέσω ισχυρών μεθοριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντα το βάρο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για γρήγορο επαναπατρισμό των προσφύγων και η Frontex να προστατεύει σωστά τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και η ανταλλαγή πληροφοριών βοηθά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Επίση υποστηρίζουμε η στατική για την αντιμετώπιση του σοβαρού εγκλήματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αντιμετωπίζουμε τι συμμορίε και τη διακίνηση όπλων, ανθρώπων, ζώων και να κατάσχονται τα παράνομα έσοδα αυτών των οργανώσεων ε, στα σύνορα ε, τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε όμω άλλα στοιχεία που παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία. Εκτό αν αυτά τα σημεία οδηγούν σε καλύτερη συνεργασία. Σίγουρα υπάρχει κάποια ηρωνία όταν ζητούμε υποχρεωτική και αμετάκλητη αλληλεγγύη αλληλεγγύη είναι κάτι που προσφέρεται, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό. Ε, βασικά, νομίζω ότι η Σουηδική Προεδρία και η ίδια η πρόταση εμπεριέχουν, εμπεριέχει πρόταση καλές ιδέες και έχει καλές ιδέες η Σουηδική Προεδρία. Δυστυχώς όμως κύριε Πρόεδρε, ε, ετοιμάζουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα με πολλά ευχολόγια και επιθυμίες και πολύ λίγα μπορούμε να πετύχουμε. Αυτό κάνουμε συνήθως. Σας ευχαριστούμε κύριε Κακό. Σας ευχαριστούμε για την Ενωτική Ευρωπαϊκή Αριστερά. Για δύο λεπτά θα λάβει τώρα τον λόγο η κυρία Έρνστ, παρακαλώ. Meine Damen und Herren. Κυρίες και κύριοι, η GUE NGL, η Ενωτική Αριστερά, δεν θα εγκρίνει αυτήν την πρόταση ψηφίσματος εδώ το ε, πρόγραμμα της Σοκχόλμης αγνοεί τις πραγματικές προκλήσεις. Επί της ουσίας, ε, μια Ευρώπη των ε, δικαίων που όμως θα ισχύουν για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως για τους αλλοδαπούς που θα ζουν σε αυτήν την Ευρώπη. Τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα ισχύουν για αυτούς. Από την άλλη τώρα πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προσυπογράψει την χάρτα ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα το οποίο χαιρετίζουμε. Από την άλλη πλευρά όμως ε, επιλέγουμε μετανάστες ως νόμιμους ή παράνομους. Η Frontex θα πρέπει να ε, τονωθεί και να ενδυναμωθεί με σημαντικό τρόπο για την καταπολέμηση λέει, των παράνομων μεταναστών. Έτσι στρεβλώνουμε την προσέγγιση των προβλημάτων της μετανάστευσης. Εδώ αποτυγχάνει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Επίσης, το μη ισορροπημένο πρόγραμμα και ο συσχετισμός ελευθερίας και της ασφάλειας. Ναι, δεν υπάρχει ε, ελευθερία χωρίς ασφάλεια, όμως ε, θα πρέπει να δούμε και το αντίστροφο. Δεν μπορούν αυτά να, να διαχωριστούν. Είναι αδιέρετα και ως ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία και, και ε, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Και, αν δεν και το θέμα των δυνατοτήτων πρέπει να εξεταστεί. Η ασφάλεια όσον αφορά τις δράσεις της αστυνομίας και τη συλλογή στοιχείων το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης ε, των ανθρώπων γίνεται κενός λόγος ε, και αχρηστεύεται. Και έτσι δεν είμαστε στη σωστή ε, διάσταση. Επιτρέψτε μου ως Γερμανίδα Ευρωβουλευτή να πω ότι 20 χρόνια μετά την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου είναι για μένα απαράδεκτο να ζω και να βιώνω πως η Ευρώπη γίνεται όλο και περισσότερο ένα οχυρό, οχυρό Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ένστα Και για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας για 1,5 λεπτό. Θα λάβει τώρα τον λόγο ο κύριος Μποργέτσιο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το έγγραφο πρόγραμμα αυτό που συζητούμε ε, βασίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά δεν δέχεται σημαντικέ τοποθετήσει τη Ιταλική κυβερνήσεω όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα. Το έγγραφο δεν αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, που, ε, επίθεση κατά του οργανωμένου εγκλήματο. Άκουσα πάρα πολλά λόγια. Θα κάνουμε τούτο το άλλο. Πολλοί αναφέρονται σε πολλέ ανησυχητικέ στοιχείε τη εγκληματικότητα. Όμω θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στι πράξει. Ε, στην ε, Ευρώπη πρέπει να κάνουμε ό,τι αυτό που κάνουμε στην Ιταλία, που είναι υπόδειγμα τη ε, καταπολέμηση, χάρη στον Υπουργό Μαρών, τη καταπολέμηση τη μαφία του οργανωμένου εγκλήματο. Δεν θέλει να κινείται η Ευρώπη προ την ίδια κατεύθυνση. Πρέπει να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό νομικό σύστημα ενιαίων. Θέλουμε να αντισταχθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη μια εγκληματικότητα που αποκτά διεθνή χαρακτήρα και κινείται άνετα μεταξύ φορολογικών παραδείσων, τραπεζών ε, και κινείται και στην αγορά κινητών και ακινήτων. Ε, και δεν δίνεται επαρκή στην. Ε, τι γίνεται με το πρόβλημα τη μετανάστευση στην Νότια Ευρώπη, όπου η συμφωνία με τη Λιβύη λειτουργεί όσον αφορά την Ιταλία και ίσω όμω να αντιμετωπιστούν κάποιε δυσκολίε εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, χρηματοδοτεί τα συστήματα επίβλεψης μέσω δορυφόρου ελέγχου των νοτιών συνόρων προς Λιβύη, εκεί που υπάρχει μεγάλη κίνηση λαθρομεταναστών. Τέλος, όσον αφορά το επεισόδιο το ρατσιστικό, κατά κάποιου εγχρώμου, ε, ε, υπήρχαν πολλοί πολλά ρατσιστικά επεισόδια που ε, γίνανε ε, κατά λευκών, εκεί που είναι θύλακες παράνομης μεταναστεύσεως ή στην ε, Νότια Αφρική την ίδια και στο βασίλειο του Μουγκάμπε. Θα πρέπει εκείνοι που μιλάνε για ρατσισμό κατά των μαύρων να θυμηθούν και ότι υπήρχαν και πολλά επεισόδια κατά των Ευρωπαίων και κατά των Λευκών τέτοια ρατσιστικά. Ευχαριστώ κύριε Μπαρκέσο για τους μη γεγραμμένους. Για ένα λεπτό δίνουμε το λόγο στον κύριο Μέλτσερ. Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η, καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης είναι σημαντικά θέματα που προκαλούν ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, ε, στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοχόλμης ε, συνεχίζεται η αρνητική στάση που υιοθέτησε το Σεπτέμβριο το Συμβούλιο. Η απλοί πολίτες, ε, μάλλον στοιχεία απλών πολιτών καταγράφονται. Ε, τούτο όμως ε, συμβαίνει στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχουν όμως διστάμενες απόψεις για το ζήτημα αυτό. Απόψεις σχετικά με, την, με το πολιτικό σορθόν σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Και τώρα προχωρούμε στους ε, άλλους ομιλητές. Ο κύριος Κασίνη για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, τις οποίες έχω την τιμή να προεδρεύω, ανέλαβα ε, το καθήκον να είμαι συγκητής για αυτό το έγγραφο μαζί με τους συγκητές Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών και της ε, Νομικής Επιτροπής. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται το 51 του Συντερικού Κανονισμού και πρέπει να πω το αποτέλεσμα, όπω το βλέπω εγώ, ήταν ικανοποιητικό, πολύ ικανοποιητικό όσον αφορά τη συνεργασία ε, μεταξύ των εισηγητών. Υπήρχαν προβλήματα και σοβαρά προβλήματα όμως όσον αφορά τον χρονισμό, το χρονοδιάγραμμα για τη συνεργασία με τους και ηγητές για την έγκαιρη μετάφραση των τροπολογιών. Είχαμε περίπου 500 Όλα αυτά οφειλόταν όμω όχι στο άρθρο 51 αυτό κάθε αυτό, αλλά περισσότερο δυσκολίε οφειλόταν στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που μα διατέθη για να ετοιμάσουμε ένα έγγραφο που θα μπορούσε να προτείνουμε στο Συμβούλιο στι 10 ε, Δεκεμβρίου. Ήταν αναπόφευκτε αυτέ οι δυσκολίε που θεόταν στον στενά χρονικά περιθώρια. Κατά λοιπά, πιστεύω ότι αντιστρόφως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία του άρθρου 51 που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Ε, το έγγραφο που παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο μας δεν μπορεί σε λίγα δευτερόλεπτα να παρουσιαστεί, που έχω στη διάθεσή μου λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά εκφράζω ικανοποίηση, διότι το σύστημα της συναποφάσεως σαν καθεστώς ε, έγινε καθεστώς συνηθισμένο της νομοθετικής διαδικασίας ε, διότι η μετανάστευση είναι θέμα ευρωπαϊκό και όχι μόνο των κρατών μελών χρειάζεται αλληλεγγύη και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο αυτή την ερμηνεία δίνουν είναι ε, ενιαίο ευρωπαϊκό πρόβλημα χρειάζεται συνεργασία των εθνικών κοινοβουλίων. Όχι σαν φύλακε που θέτουν όρια, αλλά σαν συνεργάτε επικοδομητική στην νομοθετική διαδικασία. Αναφέρθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξαιρετικά ε, σημαντικό θέμα που είναι η ψυχή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Λαμβάνοντα υπόψη ότι αυτό το έγγραφο ότι δεν έπρεπε να να μπει σε κάθε λεπτομέρεια όσον αφορά την εφαρμογή του πρόγραμματο τη Στοχόλμη, αλλά δώσει κάποιου προσανατολισμού γενικού. Από αυτή την έποψη θα πω ότι είναι θετικό το, έγγραφο και θα, ε, θα μπορέσουν ε, μετά να εξεταστούν οι λεπτομέρειε του. Ευχαριστώ κύριε Καζίνη. Δίνουμε το λόγο για δύο λεπτά, δυόμιση λεπτά ο κύριος, τον κύριο Λόπεθ Αγελάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας την Σουηδική Προεδρία, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προάγουν αυτό το πενταετές πρόγραμμα στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Τρεις επιτροπές έχουν ασχοληθεί η Επιτροπή Ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν... Για την εφαρμογή του άρθρου 51, διότι πρέπει έγκαιρα να δράσουμε για τη δημιουργία του χώρου δικαιοσύνη και ελευθερία, γνωρίζοντα ότι θα άρχιζε να ισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα, ένα μεγάλο βήμα προ τα εμπρό, Θα, ήταν, θα είναι συνομοθέτης ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασιστική σημασία στο θέμα τη διακυβερνητική μέχρι σήμερα συνεργασία. Επίση, επειδή θα αρχίσει να ισχύει η θεμελιώδης χάρτα, η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων και η εντολή επικύρωση. Ε, από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ενίσχυση δηλαδή των διαστάσεων ελευθερία και δικαιοσύνη. Η ασφάλεια δεν είναι σε αντίθεση με τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. Είναι συμπληρωματικό αγαθό και πρέπει όλα αυτά να εντάσσονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Να κατανοούμε σωστά τα δικαιώματα τη ηθαγένεια, τα δικαιώματα των πολιτών. Ένταξη, ολοκλήρωση, δικαιώμα, δικαιώματα ετούντων άσυλο, συνεργασία αστυνομική. Όλα αυτά για να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών και την προαγωγή το, της συνεργασίας, ιδιαίτερα και της δικαστικής συνεργασίας και αστυνομικής συνεργασίας για την καταπολέμηση των πραγματικών εχθρών, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Δούλεψε σκληρά το Κοινοβούλιο και βελτίωσε το έγγραφο αυτό σε σχέση με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου. Το βελτίωσε ενισχύοντας ε, την ρήτρα κατά των διακρίσεων, ιδιαίτερα κατά των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και των Υπάρχει δέσμευση κατά πολέμηση της διάστασης ε, της αδικίας και της αντική ε, διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος ε, των γυναικών. Και όλα αυτά σε σχέση με το άσυλο, όλα δείχνουν ότι το άσυλο, η μετανάστευση δεν αφορούν μόνο ένα κράτος μέλος, αλλά αφορούν τη συνεργασία όλων των κρατών μελών, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει η κατάρτιση και η εκπαίδευση των δικαστών για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να υπάρξει προσέγγιση των πλαισίων από πλευρά μα και μέσω τη αμοιβαία αναγνώριση και τη εμπιστοσύνη θα πρέπει να μπορούμε να εργαστούμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένα πραγματικό ένας πραγματικός χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Όλα αυτά νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο και έχουν νόημα. Και αύριο στην Ευρωβουλή σε σχέση με την ψήφιση της, ε, έκθεσης, της κοινοβουλευτικής έκθεσης που από κοινού η Συνταγματική Επιτροπή, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών εργαστήκαμε, θέλουμε να υπάρξει ένα σαφές μήνυμα. Είναι μεγάλη σημασία για μας έχουν ε, τα, ε, η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, των Πολιτικών Ελευθεριών. Πρέπει από κοινού να συνεργαστούμε ώστε διασυνοριακά το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία να καταπολεμηθούν και τα θύματα ιδιαίτερα της τρομοκρατίας να προστατεύονται. Οι πολίτες δεν θα κατανοούσαν αν αποτυγχάναμε. Γι' αυτό ζητώ την ευρύτερη υποστήριξη σε αυτό το σώμα για την έκθεση που αύριο θα κατατεθεί και θα υποβληθεί σε εσά για να υπερψηφιστεί. Ευχαριστώ κύριε Λόπεθ Για ένα λεπτό η κυρία Σοφία παρακαλώ. Uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα ε, στεναρά λόγια, την τοποθέτηση του Συμβουλίου και για την συνεργασία με την Ευρωβουλή. Ακόμα περισσότερο θα προτιμούσα βέβαια το Συμβούλιο να ε, ενστερνιζόταν τις συστάσεις της Ευρωβουλής, διότι διαπιστώνω ότι το Συμβούλιο συνεχίζει απλά από πλευρά του όπως και μέχρι σήμερα. Και εδώ, σε σχέση με το Κοινοβούλιο που εργάζεται για μια τοποθέτηση, δεν λαμβάνει την τοποθέτηση αυτή από το Συμβούλιο υπόψη. Τώρα, για ένα άλλο σημείο, για την κυρία Ζανίν ε, Νες που το προανέφερε. Θέλω να το υπενθυμίσω για άλλη μια φορά και ιδιαίτερα τις δύο μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Να το αναφέρω. Η ελευθερία είναι αδιέρετη και αδιαχώριστη. Δεν μπορούμε εδώ να υιοθετήσουμε κάποιες αρχές που θα ισχύουν για τους μεν ενώ για τους δε όχι. Έγινε λόγος εδώ επίσης ε, και για το ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να ασκήσουμε την επιρροή μας σε σχέση σχέση με γάμους που συνάπτονται, σε σχέση με ε, την απαγόρευση που υπήρχε έναντι ε, τέτοιων, γάμων μεταξύ μελών διαφορετικών θρησκειών ή δογμάτων ή ομολογιών. Αυτό είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν και εδώ για την αναγνώριση γάμων ε, θα πρέπει ακόμα και αν είναι του ιδίου φίλου οι δύο οι οποίοι νυμφεύονται ή παντρεύονται θα πρέπει να υπόψη, να λάβουμε υπόψη τα δικαιώματα τους και στρέφομαι ιδιαίτερα προς τους φίλους ε, που έχουμε στους σοσιαλιστές για να ληφθεί αυτό υπόψη. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και οι πολίτες οι Ευρώπη τα άτομα άσχετα ποια είναι η φυλή τους, ε, η θρησκεία τους ή η δική τους σεξουαλική επιλογή πρέπει να αναγνωρίζονται στα δικαιώματά τους πλήρως. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό επίσης για την κυρία Ταβάρες, τον κύριο Ρούι Ταβάρες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι θα ήταν ευπρόσδεκτο από πλευρά ε, του σώματος ένα πρόγραμμα Στοκχόλμης που θα ήταν εξειδικευμένο, συγκεκριμένο και θα σημείωνε πρόοδο για την Ευρώπη των πολιτών. Δυστυχώς πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά, ε, πιο πίσω από αυτούς τους στόχους που θα έπρεπε να είχαμε. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ακολουθεί μια κάποια συγκεκριμένη τάση γενικολογίας ε, αφηρημένων ενιών και προσεγγίσεων. Δεν είναι πολύ συγκεκριμένο και δεν υπάρχει δημοκρατικός κοινοβουλευτικό έλεγχος ώστε να υπάρχει υπάρχει σωστή παρέμβαση από πλευρά ε, του Κοινοβουλίου, ώστε να υπάρχει τροποποίηση και προσαρμογή εκείνων που πρέπει να προσαρμοστούν. Και αυτό αποτελεί το πρόγραμμα ε, αυτού του ελληπού προγράμματο και γενικόλογου προγράμματο τη Στοκχόλμη. Να δώσω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τι πολιτικέ μετανάστευση. Όλοι εμεί παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την ε, εφαρμογή του ΕΑΣ. Υπάρχουν πολύ λίγοι διάβλοι για το άνοιγμα νόμιμων διάβλων για τη μετανάστευση. Θα χρειαζόμαστε περισσότερο αυτή τη διάσταση. Δεν βρίσκονται όμω μέσα στο πρόγραμμα τη Στοχόλμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Για 1,5 λεπτό θα λάβει τον λόγο ο κύριο Πάτεν παρακαλώ. Το πρόγραμμα Στοκχόλμης είναι ένα τμήμα προσπάθειας δημιουργίας ενός κοινού νομικού και δικαστικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έγγραφο αναφέρεται και παραθέτω η ζωή των ανθρώπων να γίνει πιο εύκολη. Μια Ευρώπη νόμου και δικαιοσύνης. Κλείνω παράθεση. Θα ήθελα να πω το κοινό νομικό σύστημα τι έκανε για τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο Άντριο Σίμιελ, 20 χρονών άντρας από το Λονδίνο, εξεδόθη στην Ελλάδα φέτος για ανθρωποκτονία στη γλώσσα μου. Είναι τώρα σε ελληνική φυλακή και περιμένει να δικαστεί. Τα στοιχεία εναντίον του δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν τα 5 λεπτά αν τα εξέταζε ένα Βρετανικό δικαστήριο. Τα στοιχεία ε, ταυτοποίησης είναι αντιφατικά. Οι μαρτυρίες των μαρτύρων έχουν, φαίνεται σαν να έχουν ε, γραφτεί από την αστυνομία. Δύο ε, μάρτυρες είπαν ότι υποχρεώθηκαν μέσω ξυλοδαρμού να υπογράψουν δηλώσεις που αμέσως μετά ανακάλεσαν. Το εφετείο στο Λονδίνο γνώριζε πολύ καλά ότι δεν υπήρχαν πραγματικά στοιχεία κατά του κυρίου Σημείου αλλά υποχρέθηκαν να τον εκδώσουν διότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη δεν είχαν τη δύναμη να σταματήσουν την έκδοσή του. Τα Βρετανικά δικαστήρια δεν μπορούν να προστατήσουν του Βρετανού πολίτε από άδικε συλλήψει και φυλακίσεις από ξένα δικαστήρια. Είχαμε ένα πολύ καλό χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας στη Βρετανία πριν ε, μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφει την νομική προστασία που απολαμβάναμε επί στην Αγγλία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής θα καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων. Το πρόγραμμα Στοκχόλμης ίσως να αφορά τον νόμο, αλλά δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Αν οι Βρετανοί θέλουν να κρατήσουν τις ελευθερίες τους, θα πρέπει να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ένα λεπτό, ο κύριος Όβερμαϊερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Χωρίς αμφιβολία το πρόγραμμα της Στοχόλμης εμπεριέχει μια ολόκληρη σειρά θετικών πρωτοβουλειών. Η καταπολέμηση παιδικής πορνογραφίας, ε, δίκτυων ε, μέτρα για τις παράνομη μετανάστευση και τα λοιπά που υποστηρίζω. Η πρόσβαση χωρί επιφυλάξει και απεριόριστα των αστυνομικών δυνάμεων σε τράπεζε δεδομένων και στοιχείων μπορεί με αυτόν τον τρόπο να θεμητοποιείται. Εδώ όμω και την, δεν έχουμε την, ε, το κράτος ε, επόπτη και με τη διάδοση στοιχείων προ τη ΣΥΠΑ. Πρέπει να διασφαλίζουμε ότι τα στοιχεία στι τράπεζε δεδομένων δεν θα, γίνονται αντικείμενο κατάχρηση Πρέπει η προστασία τη ιδιωτική. Ε, και των προσωπικών δεδομένων να διασφαλίζεται. Ελευθερία από το κράτος, ε, σε σχέση με το κράτος και όχι ελευθερία μέσω του κράτους. Πρέπει να διασφαλίζεται αυτή η πτυχή της ελευθερίας. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να πούμε χωρίς εναρμονισμό των οικονομικών προϋποθέσεων για τη μετανάστευση δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Ακόμα η, καλύτερη διασφάλιση είναι ε, να καταστήσουμε τις πόλεις μας ε, ασφαλείς. Η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να γίνει ένα μαγαζί αυτοεξυπηρέτησης για εκείνους που επιθυμούν άσυλο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο συνάδελφος Μπουσούτιλ. E ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο τομέας της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας και το πρόγραμμα αυτό είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, το σπουδαιότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ένα παρεμφερές πρόγραμμα είναι, το, είναι η εσωτερική αγορά σε συνδυασμό με τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια για τους πολίτες. Και πώς θα φτάσουμε εκεί, μέσω του προγράμματος της Στοχόλμης Ένα πρόγραμμα εργασίας για διάστημα 5 ετών. Ένα ευρύ πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει διάφορους τομείς και πτυχές ε, ως προς την ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου προτείνει τις πολιτικές προτεραιότητες σε αυτούς τους τομείς. Παραδείγματο χάρη, μετανάστευση. Προτεραιότητά μας είναι η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Ενώ ταυτόχρονα θέλουμε μια κοινή πολιτική, ενιαία πολιτική υπέρ του ασύλου που θα εδράζεται στην πραγματική αλληλεγγύη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το οποίο οφείλει να διαδραματίσει, έναν ρόλο επικοδομητικό στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και το τελευταίο μου σχόλιο. Ασφαλώς υπάρχουν πολιτικές διαφορές εντός αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτού του σώματος. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές ομάδες και διαφορετικές απόψεις ως προς την πολιτική που ασκείται. Θα ήθελα λοιπόν, στρεφόμενος προς τη συνάδελφο Ζανίν, ε, να της πω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολιτική προτεραιότητα και για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν μονοπόλιο της φιλελεύθερης ομάδας αυτού του κοινοβουλίου. Δεν δεχόμαστε το, η αρχή της ε, μη διάκρισης είναι προνόμιο και μονοπόλιο της φιλελεύθερης ομάδας. Και εμείς πιστεύουμε στην αρχή αυτή, ενώ ταυτόχρονα πιστεύουμε στην αρχή της επικουρικότητας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τις εθνικές ευαισθησίες της Ευρωπαϊκής, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ένωση αυτή έχει οικοδομηθεί πάνω στις, στις διαφορές που υπάρχουν και όχι στην ε, απλή ενότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ είναι κάτι το οποίο υπενθυμίζω ότι μα πιέζει πολύ ο χρόνο. Έχουμε καθυστερήσει πολύ. Θα παρακαλούσα οι συνάδελφοι να τηρούν το χρονικό όριο στι παρεμβάσει του. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση όπω ε, έχει προβλεφθεί μέσα στα όρια του χρόνου. Για δυόμιση λεπτά θα λάβει τον λόγο ο συνάδελφο Μπερλουσκόνη. Ε, με συγχωρείτε, Μπερλιγκουέρ. Δύο είναι οι καινοτομίε του προγράμματος Στοχόλμη σε συγκρίση με αυτό τη χάγη, Σωστή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων ε, ασφαλεία και νομική προστασία και στον ποινικό και στον αστικό τομέα. Η ασφάλεια είναι ένα δικαίωμα. Ε, το να μην δεχτεί καμία επίθεση στον χώρο εργασία, να μπορεί να τριγυρνάει στον δρόμο χωρί να κινδυνεύει η ζωή του, να μην είναι αντικείμενο βία, ε, άμα είναι ε, γυναίκα, να μην εκτίθεται σε τρομοκρατικέ πράξει κλπ. Ε, οι, χώρε και η Ευρώπη θα πρέπει να εγγυούνται την ασφάλεια. Να εγγυούνται την ασφάλεια. Αλλά μία θα πρέπει να έχει τα χέρια ελευθερία, αυτή η ασφάλεια, όμω που βγάζει ε, την ασφάλεια από το δίκαιο. Οπότε μπορεί να ε, υπάρχουν βαρβαρότητε, όπω είναι και το Γκουαντάναμο. Είναι η πατρίδα των δικαιωμάτων η Ευρώπη. Το πρόγραμμα του Χόλμη το καθορίζει σαν ε, προστασία των ατόμων. Χρειάζεται σωστή ισορροπία μεταξύ τη της καταστολή των εγκλημάτων από τη μία πλευρά και τη κανονική ζωή των πολιτών από την άλλη. Με οικογενειακέ σχέσει, κοινωνικέ, οικονομικέ σχέσει, εργασία, ε, σπουδέ, όλα θα διευθετούνται από το αστικό δίκαιο και από τη δικαιοσύνη, την αυτή είναι η Ευρώπη του πολίτη και θα ε, πρέπει να οικοδομείται εντό των κρατών μελών και εντό των θεσμικών οργάνων τη Ένωση. Η ευρωπαϊκή κοινωνία είναι πιο ενωμένη, η κινητικότητα πιο μεγάλη από ό,τι πιστεύουμε. Η κινητικότητα τώρα πια είναι ένα δικαίωμα και τα όρια μεταξύ των κατών δεν είναι τύχη αδιαπέραστη, είναι δίκτυα μέσω των οποίων ε, ε γίνεται δίθυση της κοινωνίας καθημερινά. Η Στοκχόλμη, Στοκχόλμη είναι θεσμικός ακρογωνίος λίθος για ε, δικαστική συνεργασία με ιδέα αναγνώριση, ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ε, σε σχέση με την εθνική και κοινοτική. Ένα εθνικό, κοινοτικό, ευρωπαϊκό δίκαιο, ένας Ευρωπαίος πολίτης ένας Ευρωπαίος δικαστής, εθνικός δικαστής και κοινοτικός δικαστής. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες εμπνέονται από νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και από ευρωπαϊκούς νόμους, αλλά προέρχονται διατάξεις και από τη συμπεριφορά των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των φοιτητών, από τους εθνικούς δικαστές, και από τα ευρωπαϊκά δίκτυα εκείνο που κινούν τους δικαιοσύνη, εκ των κάτω προς τα πάνω. Και αυτό ε, θέλω να το υποστηρίξω το πρόγραμμα στο Στοχόλμη, γιατί κινείται το τρόπο. Το Κοινοβούλιο κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια μέσω αυτού του ψηφίσματο, που ε, ελπίζω να ψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία εδώ, ενιαία ψήφο, ε, κάτι για το οποίο εργαστήκαμε εντατικά. Το Συμβούλιο ε, θα πρέπει να το λάβει με σεβασμό υπόψη. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα η Λισαβόνα, αλλά είναι εκεί, παρούσα. Ε, θα πρέπει να είναι φιλόδοξο το Συμβούλιο κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει να στερνιστεί αυτά που επεξεργαστήκαμε εμείς εδώ ε, και να λάβει υπόψη τον πλούτο των διαφόρων ετοιμάτων και προτάσεων που απορρέουν από αυτό το κείμενο. Ένα λεπτό, η κυρία Λάντφορντ, παρακαλώ. Πρόεδρε, η Σουηδική Προεδρία θα πρέπει να συγχαρούμε τη Σουηδική Προεδρία για το γεγονό ότι προώθησε το θέμα των δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι θεμελιώδου σημασία ε, να, ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Η αμοιβαία αναγνώριση πραγματικά μπορεί να βασιστεί στην αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη των δικαστικών συστημάτων πράγμα που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή διότι υπάρχουν τεράστιες αδυναμίες και ο δικός μου πολίτης είναι ο Άντριος τον ε, του αρνήθηκαν τα δικαιώματά του επειδή ήταν ξένος. Ο Έλληνας ε, δικηγόρος του μίλησε για κατάχρηση εκ μέρους της αστυνομίας. Είναι πραγματικά ε, φοβερό και είναι ντροπή το, η τέτοια μεταχείριση ενός Ευρωπαίου πολίτη από κάποιον άλλον Ευρωπαίο πολίτη. Εγώ υποστηρίζω το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλλευση, ωστόσο θα πρέπει να υπάρξουν και τα δικαιώματα των πολιτών. Διαφορετικά θα έχουμε σκανδαλώδες υποθέσεις όπως αυτό του Άνδριο Σεμιά, κάτι το οποίο συμβαίνει και στη δική μου χώρα. Ευχαριστώ κυρία Λούτφορτ. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Τριανταφυλλίδη έχει το λόγο για την ανάγκη να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της ασφάλειας και της προάσπισης των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι ο πολίτης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος της Στοκχόλμης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί και εφαρμόζει μέτρα που καταλύουν το ισοζύγιο ασφάλειας δικαιωμάτων, οδηγούν στη δημιουργία σωμάτων παρακολούθησης, συλλογής παντοσίδους προσωπικών δεδομένων και παραβίασης της αξιοπρέπειας μας εφόσον όλοι μετατρεπόμαστε σε υπόπτου. Επιπρόσθετα, είναι απαράδεκτο όλοι οι μετανάστε να αντιμετωπίζονται ω εγκληματίε και πιθανοί τρομοκράτε. Εμεί διαφωνούμε με το σχέδιο ψηφίσματο γιατί θέτει τα θεμέλια για να χτίσουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανόπτικο όπου, όπω στη φυλακή που είχε σχεδιάσει ο Τζέρεμι Μπένθαμ, οι πράξει όλων παρακολουθούνται συνεχώ, χωρί να γνωρίζουν οι κρατούμενοι την έκταση αυτή τη επιτήρηση, δίνοντα του την ψευδέστηση ότι έχουν ιδιωτική ζωή. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά στη συνέχεια για τον κύριο Ταντέους Σβίφκα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δεν φοβούμε να ισχυριστώ ότι στον χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης ε, και ασφάλειας το πρόγραμμα της Στοκόλμης είναι μια πολύ φιλόδοξη πρωτοβουλία. Η καλύτερη των τελευταίων ετών, η πιο φιλόδοξη. Χαίρομαι για τις ιδέες που εμπεριέχονται σε αυτό το πρόγραμμα και η απλούστευση της ζωής των πολιτών. Η λογική εφαρμογή και εύλογη εφαρμογή του προγράμματος της Στοκόλμης εξαρτάται φυσικά από τις δομές ε, τις δικαστικές που θα δημιουργηθούν για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και να είναι αποτελεσματικό. Επίσης και το EGIS. Είναι πολύ σημαντικό και το θέμα της αμοιβαία αναγνώρισης ως θέμα αρχής για την αύξηση της εμπιστοσύνης. Χρειαζόμαστε επίσης και την τόνωση της εμπιστοσύνης στα όσα συμβαίνουν δικαστικά στις άλλες χώρες. Η καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και προσέγγιση των χωρών μας ε, και των δικαστών και των διαφορετικών νομικών πλαισίων και παραδόσεων που έχουμε. Πρέπει να προσεγγίσουμε ο ένα τον άλλο περισσότερο με ενεργό τρόπο. Πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών και βιωμάτων με ε, επισκέψεις ε, από του μεν στους δε και να έχουμε ε, κατάρτιση και επιμόρφωση μετεκπαίδευση των δικαστών και ένα εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων μα και των μαθημάτων που προσφέρουμε όταν πρόκειται για τα μαθήματα νομική και επίσης και το Aegis, το, πιλωτικό αυτό πρόγραμμα ε, η πύλη στο διαδίκτυο Aegis, ώστε διαδικτυακά ηλεκτρονικά στοιχεία να μπορούν να ανταλλάσσονται και να υπάρχουν ε, οι εγγυήσει και οι διευκολύνσεις στους πολίτες όσον αφορά το νομικό πλαίσιο και τα δικαστικά θέματα. Αυτή η δυνατότητα θα δώσει την, ε, περισσότερες δυνατότητες και σε δικηγόρους και πολίτες και για το νομικό σύστημα που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Χαίρομαι ότι αυτή η διάσταση αναφέρει προβλέφθηκε και από τον Επίτροπο Μπαρό. Χρειαζόμαστε νομοθεσία βέλτιση ανώτατη ποιότητα, πολύ αναβαθμισμένη και τη σωστή συνεργασία. Πρέπει εδώ να ασκηθεί σωστά η επιρροή μα, ώστε οι πολίτε να έχουν αποτελεσματικά μέσα στη διάθεσή του ώστε τα διαφορετικά νομικά προβλήματα στην ενιαία εσωτερική αγορά να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν σωστά. Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τι ευρωφοβίε ή του ευρωσκεπτικιστέ, δείχνοντα στου πολίτε με το πρόγραμμα τη Στοχόλμη ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν τη σωστή απάντηση στα προβλήματά τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά στη συνέχεια για την κυρία Γκουρμάη. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Στα συγχαρητήριά μου για τους συναδέλφους οι οποίοι εκπώνησαν αυτό το ψήφισμα. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, συμβάλλει ώστε να έχουμε μια πιο ασφαλή Ευρώπη ε, θα υπάρξει πρακτική συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών και δικαστικών αρχών και των αρχών των υπευθύνων για τις ε, μετανάστες και με αυτόν τον τρόπο θα επιβάλλεται το κράτος δικαίου. Ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο θέμα. Η εισαγωγή της αρχής της σύγκλησης είναι πολύ σημαντική. Είναι ένα ακόμα βήμα. Ε, δεν είναι αφαίρεση κυριαρχίας. Όλα τα στοιχεία, όλες οι πληροφορίες και η ενημέρωση θα βοηθήσουν τι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαλειτουργικότητα του συστήματος Συστήματο Πληροφόρηση Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει ώστε όλε οι υπηρεσίε να μπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία μεταξύ του. Όλα τα θέματα τη ισότητα έχουν σημασία. Το θέμα τη ισότητα των φύλων περιγράφονται στο κείμενο. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ιστορική στιγμή ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη μετά τη σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και το, μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτόν τον τρόπο γίνεται θέμα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη για το γεγονός αυτό. Ελευθερία, δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα, δημοκρατία, ισότητα και ιδιωτικότητα. Νολίζω ότι οι αξίες αυτές έχουν διαφορετικές έννοιες ανάλογα με το πολιτικό κλίμα. Το ψήφισμα όμως ε, έχει μια σωστή ισορροπία. Θα ήθελα να αναγνωρίσω ότι το, οι παράγραφοι σχετικά με την οικογένεια και τα παιδιά θα πρέπει να ενισχυθούν. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες μας χρειάζονται μια ρεαλιστική ε, πολιτική μετανάστευση επί τη βάση κοινών αρχών και κανόνων περιλαμβανομένης της αρχής της αλληλεγγύης και της διαφάνειας. Η μετανάστευση μπορεί να είναι ε, ε, και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, ε, και επίσης να βοηθήσει και τις χώρες οι οποίες έχουν μετανάστες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Ζήτα. Κατάφερε να ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν μπόρεσε η διερμηνία να σε παρακολουθήσει με αυτό το ρυθμό. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Θέλουμε να συγχαρούμε τους διερμηνεί για την επιτυχία αυτή. Δεν βλέπω να παρίσταται ο συνάδελφο Άλβαρο, που είναι ο επόμενο αγορητή. Δεν είναι στο έδρανό του, στη θέση του. Δεν ξέρω αν κάθεται αλλού σε άλλο έδρανο. Δεν τον βλέπω. Και γι' αυτό θα περάσουμε στον επόμενο αγορητή, που είναι ο κύριος Πασκάλ Γκρουνί. Η κυρία, με συγχωρείτε, διορθώνει ο πρόεδρο. Θα λάβει τον λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, κυρίε και κύριε Υπουργέ, επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν θα επαναλάβω τα βασικά στοιχεία, τα ανέφεραν οι συνάδελφοί μου όσον αφορά τα θέματα δικαιοσύνη και μετανάστευση. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι ένα ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο δεν θα μπορεί να είναι εφικτό παρά μόνο μέσω τη ενισχύσεω μια αμοιβέ εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών, που θα βελτιώσει έτσι την αρχή τη αμοιβαία αναγνώριση που είναι ακρογωνίως λήθος της Ευρώπης της δικαιοσύνης. Σημαντικές πρόοδοι έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά πολλές αδυναμίες εξακολουθούν να εφίστανται. Χαίρομαι διότι κατά διάρκεια των υπαγορευτεύσεων επί του κειμένου η συνθήκη της Σαββόνας επιτέλους επικυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να εισακουστεί σε ίση βάση όπως και το Συμβούλιο σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών ε, μια δημοκρατική νομιμότητα τελικά θα αυξηθεί προς όφελος των ε, πολιτών. Ω και εισηγήτρια του ΕΛΚ, νόμα τη Επιτροπή Αναφορών, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πάρα πολλές καταγγελίε ε, ε, καταγγελίες γίνονται στην Επιτροπή μα όσον αφορά εμπόδια για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών εντό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Θα ήθελα να επιθυμίσω το πρόβλημα που συνδέεται με βία αναγνώριση των πτυχίων, το δικαίωμα κοινωνικών παροχών και τα προβλήματα διακριτική μεταχείρισης. Αλλά όσον αφορά την αναγνώριση γάμου ατόμου του δύο φύλου, αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Ένωση θα πρέπει να σεβαστεί αυτή την εθνική αρμοδιότητα. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει πολύ γρήγορα τι κατευθύνε γραμμέ, ώστε να βοηθήσει τι αρχέ των κρατών μελών να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την κατάχρηση τη αρχή τη ελεύθερη διακίνηση. Οι πολίτε θα πρέπει να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα και να απολαμβάνουν πλήρω του δικαιώματο του αυτού ε, του εσωτερικού χώρου χωρί εσωτερικά σύνορα. Στο ψήφισμα χαίρομαι που η στρατηγική κατά των ναρκωτικών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω έχει μια θέση στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τη δικαιοσύνη. Θα ήθελα όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει περισσότερη πρωτοβουλία στον αφορά αυτό το θέμα. Γιατί η Ένωση δεν αποκτά νέο μέσα για να καταπολεμήσει το αυξανόμενο φαινόμενο αυτό που πλήττει τα παιδιά μα όλο και περισσότερο. Εκείνη είναι το μέλλον μα. Τι κάνουμε εμεί για να προστατεύσουμε τα παιδιά, να δείξουμε ρεαλισμό όσον αφορά του θεσμού μα. Αυτό περιμένουν οι συμπολίτε μα από εμά. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστούμε κυρία ο κύριος Κλοντ Μωράης, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν μια μακρά πορεία από το Τάμπερε, όπου είδαμε απλώς το περίγραμμα του χώρου ασφάλειας δικαιοσύνης και με μεγάλη συζήτηση όπου και φτάσαμε τώρα εδώ όπου Στοκχόλμη και Λισαβόνα ε, συνδυάζονται. Χρειάζεται λοιπόν εμείς να δώσουμε τη δική μας μάχη για να εξασφαλίσουμε την δικαιοσύνη και την ελευθερία και την ασφάλεια που εμείς επιδιώκουμε. Και εμείς ως ομάδα θα υπεραντιμνθούμε των προοδευτικών ε, πολιτικών μας. Και έχουμε και τη Λισαβόνα τώρα, αλλά πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας όλα τα μέλη εδώ, ανεξάρτητα από πολιτικές ομάδες, ώστε να νομοθετήσουμε μετά τα Χριστούγεννα για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ευθύνη. Και εμείς η δική μας ομάδα μετά το σκληρό έργο που έκανε η συγγητής μας έχουμε τις δικές μας προτεραιότητες και ο τομέας ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας είναι αυτός που μας ενδιαφέρει η κατάργηση των διακρίσεων. Θέλουμε μια οριζόντια οδηγία. Στείλαμε το μήνυμα στο Συμβούλιο. Ε, σχετικά με τη δικαιοσύνη. Η αμοιβαία αναγνώριση είναι πάρα πολύ σημαντική για να λειτουργήσει το ευρωπαϊκό ένταλμα ασύλου. Αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών. Για μας προοδευτική λύση σημαίνει ότι αυτοί που επιδιώκουν άσυλο, που ζητούν άσυλο να έχουν την καλύτερη εκπροσώπηση. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της ομάδας μας. Και μια πρόσθετη αξία που εμείς ε, θέτουμε είναι τα ε, εγκλήματα μίσους, τη βία εναντίον των γυναικών. Όλα αυτά δείχνουν πώς εμείς ως πολιτική ομάδα, όπως και οι άλλες πολιτικές ομάδες, μπορούν να προσθέσουν αξία στο πρόγραμμα της Στοχόλμης και για να υπάρξει νομοθεσία που θα έχει νόημα. Τελικά παίζουμε το παιχνίδι διότι για τους πολίτες μας δεν πρόκειται για παιχνίδι. Είναι να τους προσφέρουμε επιτέλους τα δικαιώματα για τα οποία αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια. Θεμελιώδη δικαιώματα, ε, ασφάλεια, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όλα αυτά θα έχουν νόημα όταν εμείς αναλάβουμε την ευθύνη και μπορέσουμε να νομοθετήσουμε. Και αυτό θα το κατορθώσουμε μέσα από το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Εμείς θα αγωνιστούμε λοιπόν για ένα τέτοιο προ... προοδευτικό πρόγραμμα της Στοχόλμης. Σας ευχαριστούμε κύριε Μουράης. Τώρα ο κύριος Καύλος Κόελιο. Δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω θερμά τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Μπαρό και την Σουηδική Προεδρία για το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Το πρόγραμμα της Στοχόλμης είναι καλά μαντάτα για όλους όσοι θέλουν να προασπιστούν την Ευρώπη Ω κάτι περισσότερο από την ενιαία εσωτερική αγορά. Η δημιουργία τη Ευρώπη των πολιτών απαιτεί έναν αυθεντικό χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Και θα πρέπει να, να ισορροπούν οι τρεις συνιστώσει αυτού του τριγώνου. Και, και οι τρεις είναι αναγκαίες. Η ασφάλεια χωρίς την ελευθερία είναι δικτατορία. Η ελευθερία χωρίς ασφάλεια είναι αναρχία και η δικαιοσύνη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς ελευθερία και χωρίς ασφάλεια. Αυτό το πρόγραμμα που είναι πενταετές αντανακλά και ε, αναπτύσσει τη φιλοδοξία του Τάμπερε και είναι σημαντικές οι συνιστώσεις αυτές. Πρέπει λοιπόν να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει ενώπιόν μας. Πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική υλοποίηση της νομοθεσίας και των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, δεν θα μας αντιμετωπίσουν ε, ως σοβαρούς πολιτικούς αν δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μια δημιουργία ενός συστήματος εισόδου-εξόδου δεν θα πρέπει να Μα ε, μας οδηγήσει στο να δράσουμε άμεσα, αλλά να περιμένουμε στο 2015. Ιδίω όσον αφορά τις ε, δράσεις ε, που είναι πιεστικές λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων. Ελπίζω ότι θα έχουμε πριν από το 2012 ένα σύστημα χωρίς ασύλου και μια πολιτική μετανάστευση με κοινή προσέγγιση και κοινέ αρχέ και σεβασμό εναντί των μεταναστών και την αποτελεσματική καταπολέμηση τη παράνομη μετανάστευση. Πρόεδρε, έχουμε πολλά να κάνουμε από κοινού για την Ευρώπη των πολιτών. Δεν έχει κανένα νόημα να χάνουμε χρόνο πια. Πρέπει να δράσουμε αποτελεσματικά. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε αρμόδιοι και να λάβουμε υπόψη και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Αυτό, αν αναμειχθούμε εμεί σε αυτές τις αρμοδιότητες, δεν είναι μόνο άχρηστο, αλλά είναι επίσης και κάτι στρεβλό. Θα πρέπει εδώ να αποφύγουμε την απομάκρυνση από το ουσιώδες. Το ουσιώδες είναι το πρόγραμμα της Στοχόλμης και πρέπει να το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κοέλιο. Και τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Χάουρεγγι. Ένα λεπτό παρακαλώ. Yeah. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να δώσω συγχαρητήρια και στη Σουηδική Προεδρία και σε όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκθεσή μας. Αλλά θα ήθελα να κάνω τρεις προειδοποίησεις πολύ σημαντικές για το μέλλον. Χωρίς νομοθετική πρωτοβουλία αν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποβάλλουν νομοθετικές πράξεις για να δώσουν σάρκα και οστά στο πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα μπορεί να αποτύχει. Δεύτερη προειδοποίηση που μου επισήμαναν οι συνάδελφοι. Το Κοινοβούλιο θα αναλάβει και νέες πρωτοβουλίες και αποστολές. Όχι μόνο εκθέσεις για απλή διαβούλευση, αλλά θα γίνει το Κοινοβούλιο συνομοθέτης Οπότε θα θα πρέπει να βρει αυτή την βλεπτή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Αυτή είναι μια νέα αποστολή και μια νέα ευθύνη για όλους τους ευρωβουλευτές. Επίσης, τρίτη προειδοποίηση για την φονταμενταλιστική εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Θα πρέπει να σεβαστούμε και τα εθνικά κοινοβούλια σίγουρα, κανένας δεν διαφωνεί με αυτό. Αλλά θα πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι μια άκαπτη και φονταμενταλιστική ερμηνεία της επικουρικότητας δεν θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε πρόοδο στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Και αν ε, οι χώρες υιοθετήσουν μια πολύ διασταλτική ερμηνεία της αρχής της επικουρικότητας, δεν θα υπάρξει κοινή νομοθεσία για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μόνικα Λουίσα Μακοβέη. Θα κάνω μια σύντομη μνήμα του τμήματο ε, τη πάταξη του οικονομικού εγκλήματο και τη διαφθορά από το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη. Δυστυχώ, στι διαπραγματεύσει ε, στι μόνιμε αντιπροσωπείε αποδυναμώθηκε κάπω το κείμενο. Για, για παράδειγμα, μιλούμε για προδιαγραφέ Γκρέκο σε ό,τι αφορά τη διαφθορά. Και είναι σημαντική η συνεργασία με τον Γκρέκο και το Συμβούλιο τη Ευρώπη, αλλά τα ευρω... οι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ πάταξη τη διαφθορά είναι πολύ ψηλότερε από τι αντίστοιχε προδιαγραφέ του Γκρέκο και του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη δεν έχει 45 μέλη και όχι 27 όπω εμεί. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω έκκληση και να παρατηρήσω το Συμβούλιο να παραμείνει σε μια ισχυρή δέσμευση υπέρ τη πάταξη τη δωροδοκία και τη διαφθορά. Χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και Μηχανισμό για να πατάξουμε την απάτη και τη διαφθορά με πολύ δυναμικό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έγγραφό μα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή τη δέσμευση και η Ευρώπη χρειάζεται μια τέτοια δέσμευση από το Συμβούλιο. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Μάικλ Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια σε όλου ε, όσοι ασχοληθούν με την έκθεση και συγχαρητήρια και προ την Σουηδική Προεδρία. Αλλάζει η, η κοινωνία. αλλάζει όχι από την μετριότητα, αλλά μέσω του θάρρου και του οράματο και αυτό ακριβώ αποδείχθηκε σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Μιλάμε για την ελευθερία την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Δύο θεμελιώδει αρχέ, ε, αλλά χωρί την ίση μεταχείριση ποτέ δεν θα έχει κανεί ελευθερία, ποτέ δεν θα έχουμε ασφάλεια και σίγουρα ποτέ δεν θα έχουμε δικαιοσύνη. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στην περίπτωση των μειονοτήτων ε, που συχνά ε, δεν εκπροσωπούνται κατά το σωστό τρόπο. Η ισότητα και η ίση μεταχείριση είναι η μόνη θεμελιώδη ακρογωνία ηλίθεια οποιασδήποτε κοινωνία και γι' αυτό Θέλω να έχουμε μια Ευρώπη στην οποία θα είμαστε όλοι ίσοι, ανεξάρτητα από την φυλή, την θρησκεία, την ηλικία, το φύλλο ή τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Μια Ευρώπη με ίση μεταχείριση, μια Ευρώπη των θεμελιωδών αξιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο συνάδελφος Ζόμπρο. Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη δίνει μια απάντηση σε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, την εξασφάλιση της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Όχι πάντα όμως, δεν δίνει πάντα ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Δεν χρειαζόμαστε ενοποίηση του ποινικού και αστικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μόνο μία εναρμόνιση και μάλιστα σε πολύ στενά προσδιορισμένους τομείς. Η Ευρώπη πάνω απ' όλα χρειάζεται αγαστή συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των δικαστικών αρχών, προκειμένου οι αποφάσεις να εφαρμόζονται σωστά και να μην μπορούν οι εγκληματίες να εκμεταλλεύονται την ελευθερία διακίνησης. Θα πρέπει επίση το πρόγραμμα της Στοχόλμης να δίνει μια σειρά εναυσμάτων και κινήτρων και σε αυτά να περιοριστεί. Θα πρέπει να παροτρύνει τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία θέματα. Καταρχήν, έχουμε την ελευθερία της διακίνησης των προσώπων. Γι' αυτό και εδώ σημαντικό είναι η συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών για τους εγκληματίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, για τα σεξουαλικά εγκλήματα που δημιουργούν απειλή για τους ε, πιο αδύναμους πολίτες ε, και τους πιο ανήμπορους που είναι τα παιδιά. Και εκεί επιστά την προσοχή μας στο πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένα μητρό των σεξουαλικών εγκλημάτων, ιδιαίτερα των πιο απειλητικών, αυτών που στρέφονται προς τα παιδιά. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε τέτοιο ε, μητρό, γιατί ε, θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για τις πιθανές ε, απειλές ε, της κοινωνίας από τέτοιους ανθρώπους που στρέφονται και έχουν θύματά τους τα παιδιά. Επίσης, τα θέματα δίμευση των περιορισιών των εγκληματιών είναι πολύ σημαντικό όργανο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Θα πρέπει έτσι με τη συνεργασία μεταξύ των κρατών να, βρεθεί, να βρεθούν τα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να διευκολύνεται η δίμευση των περιουσιακών στοιχείων των εγκληματιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τα, τα παραπτώματα και τα πλημελήματα. Μην ξεχνάτε ότι μερικές φορές η στέρηση της ελευθερίας είναι πολύ σημαντικό αγαθό και δεν θα πρέπει να επιφυλάσσεται παρά μόνο για τα σοβαρότερα εγκλήματα. Και θα πρέπει να είναι πραγματικά η ανάλογη και η δίκαιη απάντηση και να μην δίνεται για ένα απλό παράπτωμα ή ένα σήμαντο πλημέλημα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στόχο του προγράμματο Στοχόλμη θα πρέπει να είναι η ενα σημαντο πλημελημα θα ηθελα να επισημανω οτι στοχος του προγραμματο στοχολμης θα πρεπει να ειναι η καλυτερη συνεργασια μεταξύ των κρατών μελών, διαφυλάσσοντας όμως τις εθνικές ιδιαιτερότητες των ποινικών συστημάτων. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα εφαρμόσουμε τη διαδικασία Catch the Eye και θα είμαι πολύ αυστηρός ε, στην εφαρμογή της διαδικασίας. Θα δώσω το λόγο σε πέντε συναδέλφους ε, για ένα λεπτό στον καθένα και θα διακόπτω τον ομιλητή εφόσον υπερβεί αυτή την ώρα που έχει στην διάθεσή του. Θα ακολουθήσω τη σειρά των ομάδων για τους πέντε ομιλητές. Η πρώτη που θα λάβει το λόγο θα είναι η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος προς ε, μια Ευρώπη που θα είναι οι πολίτες στο κέντρο της και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Υπουργούς Άλστ και Βέλστρομ για το όραμά τους. Τέλος, μπορούμε να πούμε επιτέλους στους πολίτες στη χώρα μας, χωρίς καμία διάκριση, ότι ναι, η Ευρώπη είναι για σας και η Ευρώπη είναι μαζί σας, η Ευρώπη είμαστε εμείς. Βέβαια το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα είναι αυτό το οποίο εμείς τελικά θα διαμορφώσουμε. Ας του δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία και ας το διαμορφώσουμε κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σωστά και ας παλέψουμε για να το εφαρμόσουμε. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω διότι αποδίδεται σημασία στα παιδιά και μπορούμε επιτέλους ε, να έχουμε ενισχυμένες δράσεις για την προστασία των παιδιών συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών μεταναστών. Πιστεύω ότι είναι ε, πιο εύκολο να καταπολεμήσουμε ε, την ε, διασυνορική εγκληματικότητα κατά αυτόν τον τρόπο, τηρώντα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διακόπτει ο Πρόεδρος και Άννα Χέντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που στην ε, πλέον ε, πρόσφατη εκδοχή του προγράμματο του Στοχόλμη, τα δικαιώματα των παιδιών και τα δικαιώματα των γυναικών ε, βρίσκονται στο κέντρο, καθώ και μέτρα καταπολέμησης τη εμπορία των ανθρώπων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ψήφη του διόρθωσε σε κάποια σημεία το πρόγραμμα, αλλά λυπάμαι που τίποτα δεν αναφέρεται για τη δημιουργία μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία των παιδιών. Κάτι που πρότεινε πρόσφατα τον, το Κοινοβούλιο. Όπω είπε και ο Επίτροπο Μπαρό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα εστιάσει αρκετά στα δικαιώματα των παιδιών. Τώρα, για την εμπορία των ανθρώπων. επίση είμαι απογοητευμένη που η Προεδρία δεν ε, δημιούργησε ένα σαφή σύνδεσμο με την ε, πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια νομική βάση για να καταπολεμήσει τη βία κατά των γυναικών και να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Ο κύριος Κέλλερ. Miss Keller, please. Ms. Um, Keller, thank you. Excuse me very much. <laughs> Κυρία Κέλλερ, ναι. Δύο σημεία που θεωρεί σημαντικά η πολιτική μας ομάδα για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης Πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν κάποια σημεία που βαίνουν προ τη λάθο κατεύθυνση, διότι για μα ε, η ασφάλεια είναι ένα εργαλείο προ την επίτευξη ελευθερία. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ, μεταξύ ελευθερίας και ασφαλεία. Και όταν μιλάμε για την ενίσχυση τη Frontex, τι ακριβώ εννοείται, ε, γιατί αυτό δεν διευκρινίζεται σε καμία από τι εκδοχέ του προγράμματο τη Στοκχόλμη που εγώ διάβασα και πιστεύετε ότι θα είναι σημαντικό, θα είναι πιο σημαντικό Λοιπόν να ενισχύσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ε, της Frontex, ώστε η Frontex ε, να μην στέλνει ε, πίσω ανθρώπους που έχουν δικαίωμα να ζητούν άσυλο, κάτι το οποίο είδαμε ήδη φέτος. Θα προτιμούσα λοιπόν τέτοια μέτρα ενδυνάμωσης, γιατί πιστεύω ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα πρέπει να υπηρετεί όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο λίγους από αυτούς. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Χιμένεθ Βεσερίγη. Είναι αναφίβολο τη σήμερα ημέρα ότι η δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση τάσεται υπέρ τη καταπολέμησης τρομοκρατία και χάρη στο πρόγραμμα της ε, κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα στο χώρο τη ελευθερία ασφάλεια και δικαιοσύνη, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό όμω ο αγώνα θα πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Ήρθε η ώρα και με τη δυνατότητα που μα προσφέρει και η συνθήκη τη Λισαβόνα να εναρμονίσουμε τι εθνικέ νομοθεσίε προ την κατεύθυνση τη μη παραγραφή των εγκλημάτων τη Τρομοκρατία που θα πρέπει να θεωρηθούν ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα μπορεί κανένας να προασπίζεται την τρομοκρατία όπως συμβαίνει μερικές φορές, γιατί είναι ανεπανόρθωτες οι ζημιές ε, και οι βλάβες των ε, θυμάτων της τρομοκρατίας που μερικές φορές βλέπουν την εξήμνηση των ε, θητών ενώ οι ίδιοι ζουν την οδύνη τους σιωπηρά. Επίσης ε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε την, ε, το, το καθήκον που έχουμε να θυμόμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Το λόγο κυρία Σιλβίκη Γιώμ. Πολλά από αυτά που ακούστηκαν σήμερα για το πρόγραμμα Στοκόλμη είναι πολύ σημαντικά. Ε, το να βρούμε μια ευρεία συνένεση και το να είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα είναι πολύ θετικά. Ε, Ούτω ή άλλω αυτά θα λέει και το αυριανό ψήφισμα που θα ψηφίσουμε. Ε, λυπάμαι που δεν αναφέρονται καθόλου οι μη κοινοτικοί κάτοικοι και οι ασθενεί. Ε, επίσης θα πρέπει να υιοθετηθεί η οδηγία για τη μη διάκριση ε, και η οδηγία για, τις, για όλες τις οικογένειες. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια για την οικογενική επανένωση και για την επανένωση των ε, ασυνόδευτων ανηλίκων με τους γονείς τους. Η ύπαρξη λοιπόν συγκεκριμένων στόχων για τους πολίτες ο σεβασμός του νέου ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, η συναπόφαση είναι μια προσθέμενη αξία, η εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, και η ορατότητα από τους πολίτες και από τη νέα γενιά του προγράμματος Στοκχόλμης, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υιοθετήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Catch the Eye. Και λυπούμε που δεν μπόρεσαν να λάβουν το λόγο και άλλοι 10-12 συνάδελφοι που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον. Αλλά ο κανονισμός μας δεσμεύει να είμαστε αυστηροί. Θα δώσω τώρα το λόγο για να απαντήσουν στους ομιλητές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση στην ε, Υπουργό Μπεατρίς Άσκ, εκ μέρους Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και Ευχαριστώ όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση για τις απόψεις που εξέφρασαν. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την υψηλή προσήλωση των Ευρωβουλευτών σε τόσο αυτά σημαντικά θέματα του προγράμματος Στοκχόλμης. Κάποιος χαρακτήρισε το πρόγραμμα φιλόδοξο και χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό, γιατί πραγματικά ήταν πολύ φιλόδοξο το έργο μας. Αλλά είναι ναι, ταυτόχρονα και ρεαλιστικό, γιατί προσπαθήσαμε να δώσουμε στο όραμά μας ε, μια ρεαλιστική προσέγγιση και να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση για τους ε, συμπολίτες μας. Ακούγοντας όμως τις παρεμβάσεις, ε, διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλη αποδοχή του σχεδίου προγράμματος της Στοκχόλμης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του τύπου, από τη σημερινή συζήτηση δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση, γιατί μερικοί μιλούσαν για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, αλλά ουσιαστικά αναφέροντας το σχέδιο ψηφίσματος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή αναφέροντας την ε, γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του προγράμματος Στοχόλμης που ήταν πρόταση της Σουηδικής Προεδρίας. Κάποιο είπε στην αρχή της συζήτηση, γιατί να συζητούμε τώρα ένα σχέδιο ψηφίσματος όταν έχει υποβληθεί νέο σχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση της ε, διαδικασίας συζήτησης και τα πράγματα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή και ίσως στην Παρασκευή ή το Σαββατοκύριακο θα υποβληθεί ένα νέο σχέδιο. Κάποιος είπε ότι συζητάτε τώρα το προηγούμενο έγγραφο. Αλλά αν δείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου, βλέπετε ότι υπάρχει ενημέρωση και η παρουσίαση των τελευταίων εκδοχών του σχεδίου. Βλέπετε ότι λαμβάνονται υπόψη συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και χάρη στις ε, προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροποποιείται και το πρόγραμμα της ε, Προεδρίας, γιατί για μας η διαφάνεια και το άνοιγμα είναι πολύ σημαντικές αρχές. Γι' αυτό έγιναν τόσε πολλέ συζητήσεις για το πρόγραμμα αυτό. Και αν στο παρελθόν ε, δεν καταφέρατε να λάβετε το λόγο ή δεν μπορέσατε σήμερα να εκφράσετε τη γνώμη σας στη συζήτηση, μπορείτε να στείλετε ένα mail είτε σε μένα είτε στον κύριο Μπίλστρομ με τις προτάσεις σας και τις υποδείξεις για να ληφθούν υπόψη και οι δικές σας ε, απόψεις γιατί επαναλαμβάνω η διαφάνεια είναι ιδιαίτερα προσφυλή στη Σουηδική Προεδρία. Και περιμένουμε ανυπομονησία το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί διαπιστώνω ότι υπάρχει ενθουσιασμός για το πρόγραμμα της Στοχόλμης και μεγάλη υποστήριξη. Μάλιστα δώσατε έμφαση και σε ορισμένα σημεία του ψηφίσματός σα που θα τα λάβουμε υπόψη και στη δική μας πρόταση. Βέβαια ανέκυψαν και κάποια πολιτικά ζητήματα που θα ήθελα να αναφέρω. Δύο ευρωβουλευτές μίλησαν και έδωσαν συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς ε, κάποιες ε, χώρες επηρεάζονται από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Και είπαν ότι ίσως είναι δυσανάλογο σε ορισμένα σημεία το πρόγραμμα αυτό. Ίσως δεν ε, υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη στα νομικά συστήματα, τα δικαιϊκά συστήματα των κρατών μελών. Είναι σαν να λέει ο καθένα στου πολίτε του καλύτερα να παραμείνετε στην πατρίδα σα γιατί το δικό μα δικαϊκό σύστημα είναι το καλύτερο. Αλλά οι πολίτε θα συνεχίσουν να παίρνουν τα σύνορα, θα εκμεταλλεύονται την ελεύθερη διακίνηση για να αξιοποιήσουν και τα ωφέλη τη εσωτερική αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιώσουμε τα δικονομικά δικαιώματα των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό το στόχο έχει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη βελτίωση των δικονομικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Για να εξασφαλίσουμε σε όλους που είτε είναι θύματα μιας εγκληματικής πράξης είτε κατηγορούμενος μιας τέτοιας πράξης να δικαιούται μετάφραση των δικογράφων υπηρεσίες διερμήνειας στη δίκη. Βέβαια, αυτό περιλαμβάνεται και στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά τώρα θα εφαρμοστεί και εμπράκτος. Η κυρία Μακοβέη μίλησε για τα οικονομικά εγκλήματα και την πάταξη της διαφθοράς και θεώρησε κάπως χαλαρό και επικές το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ως προς αυτό το σημείο. Νομίζω ότι είμαστε σαφείς. Αναφέραμε τον Γκρέκο, τις προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά δεν είπαμε ότι θα περιοριστούμε σε αυτές ε, τις ε, σχετικά μικρές προσδοκίες είπαμε ότι θα έχουμε στενότερη συνεργασία με αυτό το σημαντικό ίδρυμα. Γιατί αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα, χρειαζόμαστε και χρηματοδότηση αυτών των προσπαθειών. Πολλοί αναφέρθηκαν και στην επικουρικότητα. Πιστεύω ότι η πρόταση που εξετάζουμε είναι πολύ σαφής ως προς την αρχή της επικουρικότητας. Λέμε ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία σε νομικά θέματα θα πρέπει να επιφέρει προστιθέμενη αξία. Ό,τι κάνουν καλύτερα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παραμείνει σε εθνικό επίπεδο. Όταν όμω χρειάζεται διασυνοριακή συνεργασία, εκεί είναι που θα χρησιμοποιήσουμε τα κοινοτικά όργανα. Δεν νομίζω ότι καταπατούμε ή σφετεριζόμαστε τα δικαιώματα των κρατών μελών. Απλώ όπου μπορούμε να συμβάλλουμε και να επιφέρουμε προστιθέμενη αξία προ όφελο των πολιτών, το επιδιώκουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, προφύλαξη τη ακαιρεότητα και την προστασία των δεδομένων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αν δεν κάνω λάθο, ο Μάριο Μποργέζιο αναφέρθηκε στο σημείο αυτό και είπε ότι υπήρξαν σοβαρές αμφιβολίες που ε, πηγάζουν από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης για το θέμα της προστασίας των δεδομένων και μίλησε για μεγάλες ε, βάσεις δεδομένων ή παρακολούθησης γίνεται ένας παραλληλισμός με το δικό μας έργο και την κατάσταση ε, στις πρώην κομμουνιστικές χώρες και τα συστήματα που εφάρμοζαν τότε. Τέτοιου είδους ε, παρομοιώσεις και επιχειρήματα είναι τελείως αναδαφικά και αβάσιμα. Στην Ανατολική Δημοκρατία δεν υπήρχε, στην Ανατολική Γερμανία δεν υπήρχε καμία προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων ή ε, καμία δημοκρατία. Άλλωστε εδώ στηριζόμαστε στην συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ενισχύουμε τους κανόνες ε, για τα προσωπικά δεδομένα, για την προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών. Σε πολλές ε, περιπτώσεις και σε πολλούς τομείς κατοχυρώσαμε αυτά τα δικαιώματα και ενισχύσαμε την προστασία τους. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της μεθοδικής και αποτελεσματικής ανταλλαγής των πληροφοριών με την ισχυρότερη προστασία των προσωπικών δεδομένων για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα στη διαχείριση των δεδομένων και η ασφάλεια των δεδομένων. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να μελετήσετε προσεκτικά τα σχετικά εδάφια του προγράμματος Στοχόλμης, γιατί εκεί μας επένεσε και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής που ασχολείται με θέματα προστασίας δεδομένων. Σε ένα άλλο θέμα που είμαστε ιδιαίτερα πρακτικοί και συγκεκριμένοι είναι ακριβώς αυτό γιατί είπατε ότι μας πιέζει ο χρόνος και στο μέλλον ε, θα σφίξουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα ως προς την πίεση του χρόνου. Γι' αυτό και θα πρέπει να συνεργαστούμε στο επόμενο στάδιο που θα είναι η εφαρμογή του προγράμματος Στοχόλμης και η θέση ισχύ των ε, διαφόρων πτυχών του προγράμματος. Εκεί έχουμε και πολλές προκλήσεις αλλά και πολλές ευκαιρίες που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ και αν θέλετε να έρθετε σε επαφή με την ε, Σουηδική Προεδρία τις επόμενες μέρες σας παραπέμπω στο διαδικτύο και στην ιστοσελίδα μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την πολύ διεξοδική σας απάντηση. Εκ μέρους του Συμβουλίου και πάλι θα δώσω το λόγο στον Υπουργό Τομπίας Μπίλστρομ. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, συμφωνώ πλήρως με τα όσα είπε η κυρία Άσκα για τα συμπεράσματα του προγράμματος και σας ευχαριστώ για τις απόψεις που διατυπώσατε σήμερα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους Προέδρους των τριών Επιτροπών συνταγματικών υποθέσεων, νομικών υποθέσεων και δημοσίων ελευθεριών για τα σχόλιά τους. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, η στάση τους δείχνει ότι πραγματικά αντιμετωπίζουν και προσεγγίζουν το θέμα με ευθύνη. Και νομίζω ότι είμαστε περήφανοι που συνεργαστήκαμε. Θα ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία για όλους τους σημαντικούς τομείς του προγράμματος. Και ο κύριος Μπουσουτήλ, όταν πήρε το λόγο, έκανε μια σύγκριση με το μέγεθος εσωτερικής αγοράς. Νομίζω ότι εύλογη είναι αυτή η σύγκριση. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό και είναι συγκρίσιμο τελικά με την εσωτερική αγορά. Κάτι που ακούσαμε για αυτό το πρόγραμμα είναι η αλληλεγγύη. Το ακούσαμε πλειστάκι. Όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των τρίτων χωρών. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα θέλαμε να περάσει μέσω του προγράμματος Στοκχόλμης. Όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, θεωρούμε ότι αυτό το περίπλοκο θέμα, οι περίπλοκες αυτές ερωτήσεις, ε, χρειάζονται βιώσιμες ε, και σοβαρές απαντήσεις. Γι' αυτό θέσαμε την αλληλεγγύη ως ε, θεμελιώδη αρχή σε όλα τα στοιχεία του προγράμματος της Στοκχόλμη και όχι σε μία παράγραφο μόνο. Και νομίζω ότι η όλη προσέγγιση στη μετανάστευση θα πρέπει να είναι ε, ο ακρογωνιαίος λήθος του προγράμματος της ε, Στοκχόλμη. Αυτό νομίζω ε, το ανέφερε και ένας από τους βουλευτές. Η Frontex δεν είναι η μόνη απάντηση στα προβλήματα και στα θέματα της μετανάστευσης η Frontex είναι ένας τρόπος για να συντονίσουμε τον έλεγχο των συνόρων των κρατών μελών. Αλλά η Frontex δεν έχει καμία εντολή σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την ακτοφυλακή. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε νομίζω ότι χρειάζεται πολλαπλών απαντήσεων. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών προέλευσης και των χωρών διέλευσης Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε βοήθεια και αναπτυξιακή αρρωγή. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον θα εμπλακεί πάρα πολύ, μια και η συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί όσον ούπο ισχύει. Ο δημοκρατικός έλεγχος θα αυξηθεί επομένω εξαιτία αυτών. Ε, σημαντικό βέβαια είναι να τονίσουμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα επιφέρει και τεράστιες αλλαγές. Οι μεγάλες αυτές αλλαγές σημαίνουν ότι ο τρόπος που νομοθετούμε στο μέλλον και αυτό θα αλλάξει. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει περισσότερη ισχύ, περισσότερο, περισσότερη εξουσία σε αυτό το τομέα. Ε, η κυρία Κέλλερα εξέφρασε κάποιες ανησυχίες εδώ, αλλά νομίζω ότι στην πραγματικότητα κινούμαστε προς μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο προς τον τομέα αυτό. Ε, συμπερασματικά και για να μην μακρηγορώ, Πρόεδρε, συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Άσκ, ότι αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να μας στείλετε email ή να επισκεφτείτε στο σελίδα μας. Ευχαριστούμε κύριε Μπίλστρομ. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με την ε, παρέμβαση του Επιτρόπου Μπαρό που θα έχει και το τελικό λόγο σε αυτή τη τόσο πλούσια συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι τρεις επιτροπές έκαναν εξαίρετη δουλειά. Η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων με τον κύριο Κασίνη που είναι παρόν, η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών με τον κύριο Λόπες Αγγιλάρ και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επίσης. Είναι μια δουλειά η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από τις τρεις επιτροπές και θα μας βοηθήσει και εμάς αλλά και τη Σουηδική Προεδρία να, δώσουμε, να οριστικοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ο, όπως είπε και ο κύριος Σιμών Μπουσουτήλ, η πολιτική αγορά, αλλά δεν διαθέτουν ένα χώρο δικαίου, ασφάλειας και ελευθερίας. Παρότι χάρη στον χώρο του Σέγγεν η ελευθερία της κυκλοφορίας είναι τώρα εξασφαλισμένη. Θα πρέπει να κρατήσουμε το όφελο. Θέλω να σας τονίσω ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εναντίον των καταχρήσεων έχουν ήδη δημοσιευθεί. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το κείμενο μου φαίνεται αρκετά ισορροπημένο. Αφού άκουσα τις διάφορες υποδείξεις και σχόλια, θεωρώ ότι αυτό το κείμενο ε, έχει φτάσει τώρα σε μια κάποια ισορροπία. Ε, να μην ξεχνάμε ότι εγγράφουμε τη Στοκχόλμη μέσα σε ένα κόσμο, μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η οργανωμένη εγκληματικότητα και η κυβέρνο εγκληματικότητα αναπτύσσεται, η τρομοκρατία αυξάνεται και φυσικά εμείς θα πρέπει να ανασκουμποθούμε. Και νομίζω ότι εδώ η Ευρώπη μπορεί να επιφέρει θέμενη αξία. Επίσης, όλο και περισσότερο σε αυτό το χώρο, τον δικαστικό, των πολιτών, έχουμε ε, ζευγάρια που αποτελούνται από ε, συντρόφους διαφορετικής εθνικότητας. Θα πρέπει λοιπόν τα ζευγάρια αυτά ε, να χρησιμοποιήσουν και να επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους στα διάφορα κράτη που ζουν και διαβιούν. Επίσης θα προχωρήσουμε στις δικονομικές εγγύησεις, όπως είπε και η Μπεατρίς Σάσκ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του προγράμματος του Στοκχόλμης στα δικονομικά θέματα. Αναφέρεται το παράδειγμα ενός πολίτη Βρετανού που βρίσκεται στην Ελλάδα. Αν υπήρχαν ελάχιστες διαδικασίες θα διευκολύνονταν τα πράγματα. Να πω και κάτι που είπε ο κύριος Κοέγιο. Ε, από το Τάμπερε μέχρι σήμερα διατρέξαμε μια τεράστια απόσταση. Επίσης, δεν μπορούμε να, να δεχτούμε τη φράση του φρουρίου. Είναι θέμα ισορροπίας μιας μεταναστευτικής ε, ευρωπαϊκής πολιτικής, γιατί αν αρνηθούμε την ε, λαθρομετανάστευση, το κάνουμε γιατί υπάρχει από πίσω το λαθρεμπόριο και το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Από την άλλη όμως είναι αλήθεια ότι καταφέραμε να παρουσιάσουμε μια πολιτική ασύλου που είναι στο ύψος των ευρωπαϊκών αξιών και της γενεοδορίας μας. Φυσικά δεν απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις, Πρόεδρε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Θα ήθελα να σας πω μονάχα ότι αυτό το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, όπως είπε και η Μπεατρίς Άσκ, είναι πραγματικά ρεαλιστικό και θα οδηγήσει σε ένα σχέδιο δράσης που η Ισπανική Προεδρία θα υλοποιήσει με τη σειρά τη και εσείς κυρίες και κύριοι βουλευτές θα είσαστε πραγματικοί συνομοθέτες θα είσαστε ένα σημαντικό εργαλείο για να προχωρήσει αυτός ο χώρος ε, δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Κάτι που επιθυμούν και οι πολίτες. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για όλα όσα έχει κάνει ήδη και για όσα θα κάνει στο μέλλον. Μια και θα εμπλακεί 100% σε αυτά τα νομοθετήματα για το χώρο δικαίου και ασφάλειας. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έχουμε λάβει ε, μια πρόταση συζήτηση. Β70155 του 2009 από τις Επιτροπές Πολιτικών Ελευθεριών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Σταγματικών Υποθέσεων. Η ψηφοφορία του ψηφίσματος αυτού θα λάβει χώρα αύριο το μεσημέρι από τις 12 και μετά. Χαίρετε αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι θα προεδρεύσω στα Ουγγρικά. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης που είναι δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις κοινέ επιχειρήσεις απομάκρυση.